Καλημέρα σα. Θα ξεκινήσουμε τι εργασίε μα. Στο πρώτο σημείο έχουμε την έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχουν παρατηρήσει, οπότε εγκρίνεται. Από πλευρά μου δεν έχω καμία ανακοίνωση. Σημείο 3 λοιπόν τραποποίηση του κανονισμού περί του καταλόγου τρίτων χωρών, οι υπηκόοι των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση θεώρηση για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και του καταλόγου τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. Ο, ο υπεύθυνο για τη γνωμοδότηση είναι ο συνάδελφο Αντρέη Κόβατσεφ του ΕΛΚΑ, τον καλωσορίζουμε. Και επί τη ουσία αρμόδιο είναι ο κύριο Αγκουστίν Δία Δεμέρα Γκαρσία Το λόγο έχει ο εισηγητής. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλου του συνάδελφου για τι προτάσει του, τι οποίε έλαβα υπόψη στην σύνταξη τη μου και στην αιτιολόγηση τη γνωμοδότησή μου. Μετά από δεκαετίε ένταση, το πολιτικό ε, κλίμα ανάμεσα στην Αλβανία και την Κίνα είναι εξαιρετικά θετικό και αυτό αποδεικνύεται μέσω της θέσπισης άμεσων πτήσεων, ε, απευθείας πτήσεων ανάμεσα στις δύο χώρες καθώς και της, ε, της συμφωνίας πλαισίου για την οικονομική συνεργασία. Οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ταϊβάνου επίσης έχουν ε, παίρνουν μια πολύ θετική τάση. Έχουμε πολύ μεγάλες ανταλλαγές επιχειρηματικές αλλά και ακαδημαϊκού επίπεδου. Έχουμε τη συνεργασία της Ταϊβάν με την Ιαπωνία και την Νότιο Κορέα. Το κατακεφαλήν εισόδημα είναι συγκρίσιμο με τη στάνταρ του ΩΣΑ. Μπορούμε να πούμε ότι το ΑΕΠ κατά κεφαλήν είναι 33.000 αμερικανικά δολάρια. Με τη βάση αυτών των τάσεων η Κομισιόν προτείνει εξαίρεση από την υποχρέωση θεώρησης ε, των υπηκών αυτών των χωρών. Η δική μου γνωμοδότηση είναι θετική. Μόνο η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Κύπρος δεν χρειάζονται, ε, είναι υποχρεούνται στην έκδοση βίζας για να επισκεφθούν την Ταϊβάν. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία ήδη έχουν άρει την απέτηση έκδοσης ε, ΒΙΖΑ για τους ε, κατόχους ταϊβανικών ε, διαβατηρίων. Η πρόταση της Κομισιόν συμπεριλαμβάνει επίσης εξαίρεση αποθεώρηση για τη μικροσκοπικό αρχιπέλαγο των βορείων νήσων Μαριάνες. Είναι ένα μικρό αρχιπέλαγος με 90.000 κατοίκους που όλοι κατέχουν διαβατήριο των ΙΠΑ. Ήθελα να κάνω το τελευταίο σχόλιο και μια μικρή αλλαγή στο κείμενο που έχει κυκλοφορήσει νωρίτερα να μπει μια φράση στην τρίτη παράγραφο που θα λέει το εξή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των Ταϊβανών στις, της Ταϊβάν στις διεθνείς ε, οργανισμούς. Αυτό θα ενισχύσει την επιχειρηματολογία της νομοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της ε, ε, προσκολούνται στην ε, πολιτική στην, στην πολιτική της μίας Κίνας, της μίας και ενωμένης Κίνας. <coughs> Δεν έχουν υποβληθεί τροπολογίες στην, στις προθεσμίες και νομίζω ότι θα μπορέσετε κι εσείς να εγκρίνετε αυτή τη γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ήσασταν τόσο πιστικός που δεν έχουν υποβληθεί οι τροπολογίες. Και η ψηφοφορία θα γίνει απόψε. Περνάμε στο σημείο 5. Λείπει όμως η συγγετρία δυστυχώς. Η κυρία Μούνης Ντε Ουρκίζα. Παρακαλώ. Ναι. Είμαι ο σκιώδης για το θέμα της ε, άρσης της υποχρέωσης θεώρησης για τους κατόχους ε, ταϊβανικών διαβατηρίων. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που μας είπε ο εισηγητής ότι οι κινέζικες αρχές δεν εξέφρασαν μέχρι στιγμής αντιρρήσεις ε, επί της προτάσεως, οπότε δεν θα υπάρξουν ούτε διπλωματικές ε, επιπλοκές. Επίσης, περιμένουμε να απαιτείται ε, θεώρηση για τους πολίτες Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Κύπρου και νομίζω ότι αυτό θα καλό θα ήταν να διορθωθεί το συντομότερο δυνατό και πριν τη λήψη της δικής μας απόφασης. Ε, Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι πρέπει να διακόψουμε την αναμονή της εισηγήτριας. Seduta sospesa quindi. Διακοπή τη συνεδρίασης. Diciamo 10 minuti. 10 minuti di sospensione più o meno dovremmo. λεπτά διάλειμμα για να έρθει και η συνάδελφος. Bene, colleghi, riprendiamo i lavori. Siamo al punto 5, accordo istituzionale. Σημείο 5. Διοργανική συμφωνία για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα. Με την έναρξη ισχύω τη Λισαβόνα είναι απαραίτητο να προβούμε σε αναθεώρηση τη Διοργανική Συμφωνία όσον αφορά την ε, δημοσιονομική επιθελτότητα που ανέρχεται στο 2006. Ε, αυτή η συμφωνία συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένες διατάξεις όσον αφορά την ΚΕΠΑ και ε, την ενημέρωση του Κοινοβουλίου σε σχέση με τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Γι' αυτό το λόγο η ανανέωση της συμφωνίας είναι μεγάλο ενδιαφέροντος για την Επιτροπή μας. Το νέο κείμενο που προτείνει η Κομισιόν αφήνει σχεδόν απαράλλακτε τι διατάξει που αφορούν την ΚΕΠΑ παρά τις ε, καινοτομίε τη συνθήκη της Λισαβόνα. Η συγγήτρια, η κυρία Μουνής, έχει αναλύσει το κείμενο που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προτείνει μια σειρά από τροπολογίε, ε, ώστε να προστατευτούν περισσότερο οι πολιτικέ και δημοσιονομικέ αρμοδιότητε του Κοινοβουλίου στον τομέα τη ΚΕΠΑ. Δίνω λοιπόν το λόγο αμέσω στην κυρία Μουνής. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντω, η συνθήκη τη Λισαβόνα προβλέπει νέε διαδικασίες, νέα θεσμικά όργανα, αλλά και νέες αρμοδιότητες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε δημοσιονομικά θέματα και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και κοινή πολιτική ασφάλειας. Οπότε είναι σκόπιμο να γίνει μια αναθεώρηση τη διοργανικής Συμφωνία για θέματα δημοσιονομική πειθαρχία μία διοργανική συμφωνία που συνήθι το 2006, οπότε καλό είναι να επικαιροποιηθεί. Το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όμως προτείνει μόνο κάποιες ε, τεχνικές αλλαγές. Στη δική μου γνωμοδότηση προτείνω μία σειρά τροποποιήσεων για να προσαρμόσουμε τη διοργανική συμφωνία στη νέα κατάσταση, δηλαδή και στο γράμμα, αλλά πρώτα απ' όλα στο πνεύμα της ε, νέας συνθήκης της Λισαβόνας. Η γνωμοδότησή μου προβλέπει και συγκεκριμένες συστάσεις, αλλά και μια σειρά τροπολογιών στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό που ουσιαστικά ζητάμε από τις γραπτές ε, συστάσεις της γνωμοδότησης και θα το συζητήσουμε είναι περισσότερη διαφάνεια ενημέρωση και τακτικές διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την ε, δημοσιονομική διαδικασία. Η ύπατη εκπρόσωπος θα πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας και από τη δήλωσή της ε, πολιτικής ευθύνης, ενημερώνοντας σωστά το Κοινοβούλιο για τις διάφορες αποστολές ε, και ΠΑ και τις ε, επιπτώσεις του στον προϋπολογισμό και επίσης θα πρέπει εκ των προτέρων να μας ενημερώνει για τις εντολές και τις στρατηγικές στα θέματα κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δίνει τη γνώμη του πριν την ε, έναρξη των αποστολών και πά και θα πρέπει να μπορεί να ελέγχει τις ε, μη στρατιωτικές αποστολές που εμπίπτουν στα πλαίσια της ΚΕΠΑ ένα τμήμα των συστάσεων που υποβάλλω στη γνωμοδότησή μου στόχο έχουν την ε, βελτίωση και την ενίσχυση των ε, ήδη προβλεπόμενων ε, συναντήσεων διαβούλευσης που λαμβάνουν χώρα μεταξύ της Επιτροπής μας και, της Προεδρίας, της, και του Προεδρίου της Πολιτικής Ασφάλειας. Προτείνουμε πέντε τέτοιες συναντήσεις το χρόνο εκτός και αν υπάρχουν φυσικά πρόβλεπτες καταστάσεις με δημοσιονομικές επιπτώσεις. Επίσης, στις ε, κοινέ αυτές συνεδριάσεις προτείνω να συμμετέχει και το Διευρυμένο Προεδρείο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών και υψηλόβαθμων ε, αξιωματούχων της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ανάλογα με το περιεχόμενο που θα έχουν οι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίση, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται για το αποτέλεσμα των αποστολών ώστε να μπορεί στο μέλλον να βελτιώνει τον προγραμματισμό τους και τη διαχείρισή τους. Στη γνωμοδότησή μου προτείνω ένα νέο σημείο αφετηρίας ε, ως προς τη διαφάνεια για τον προϋπολογισμό της ΚΕΠΑ και προβλέ... προτείνω ενημέρωση και τακτικέ διαβουλεύσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι καλό θα είναι να ενημερωνόμαστε και για τη χρηματοδότηση επίγουσών πρωτοβουλειών σε ό,τι αφορά θέματα ασφάλειας και άμυνας. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στέλνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το αποτέλεσμα των ελέγχων για δράσεις και αποφάσεις σε θέματα ΚΕΠΑ. ΚΕΠΑ. Αυτό είναι το περιεχόμενο σε γενικές γραμμές της γνωμοδότησής μου. Ελπίζω να μη διαφωνήσετε, γιατί ουσιαστικά προσπαθώ μέσω της Επιτροπής Εξωτερικών να επαναφέρω το Κοινοβούλιο στην θέση που του αξίζει με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας και τις νέες αρμοδιότητες που προβλέπει αυτή για τον προϋπολογισμό και για την ΚΕΠΑ. Έχουμε προβλέψει και προθεσμοί για τις τροπολογίες. Ευελπιστώ πάντως ότι θα συμφωνήσετε με το γενικό προσανατολισμό της έκθεσης, της Γραμματότητας μάλλον, και θα την υποστηρίξετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφε μου, να θυμίσω ότι η προθεσμία για υποβολή του υπολογιών είναι η 7η Οκτωβρίου και η ψηφοφορία θα είναι στις 27 Οκτωβρίου. Προβλέπεται η ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Νοέμβριο. Οπότε μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Πρώτος είναι ο κ. Λέζινγκ. Η κυρία, συγγνώμη, Λέζινγκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για την ομοδότησή σας. Θα ήθελα να είμαι σύντομη και η ομάδα μου και εγώ χαιρετίζουμε την ε, τροπολογία σας για την ε, δια, δια, διοργανική συνεργασία, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή, έλεγχος και διαφάνεια από το Κοινοβούλιο για τον έλεγχο του προπολογισμού. Σε πολλά άλλα σημεία βεβαίω έχουμε αρκετά προβλήματα, ειδικά σε ό,τι αφορά την, την αποθεματοποίηση των ε, κονδυλίων για την κοινή ε, πολιτική, και την εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνα. Ε, θεωρούμε ότι εκεί θα πρέπει να ακολουθήσουμε άλλη γραμμή. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει η Ευρώπη να είναι μια, ένας φορέας που παράγει ειρήνη και πολιτισμό και ότι δεν θα πρέπει να συνδεθεί με στρατιωτικές ή πολιτικές ε, ε επιχειρήσεις. Επίσης είμαστε της άποψης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω οικονομικού και πολιτικού οικονομικών και πολιτικών διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να προχωρήσει. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί ε, φιλελεύθερα μέσα για να μειώσει την... Ε, ε, το περιθώριο έλλειμμων που έχουν άλλες χώρες. Προς το παρόν, στην εξωτερική πολιτική που ασκούμε, δεν βλέπουμε καμία βελτίωση ή καμία μεγαλύτερη νομιμοποίηση των ε, στρατιωτικών επιχειρήσεων. έτσι ώστε να δικαιολογείται ας πούμε η χρήση τους για, την, για τον εκδημοκρατισμό. Ε, δεν νομίζουμε ότι αλλάζει ο χαρακτήρας αυτών των ε, επιχειρήσεων, οπότε πιστεύουμε ότι τα ε, κονδύλια αυτά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για, για ε, στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά μόνο για ε, ειρηνικές ή ειρηνοποιητικές ε, επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλοι συνάδελφοι θέλουν το λόγο. Κανείς. Α, παρακαλώ κυρία Νέιτς. Meneer de voorzitter, waarde collega's, ik zou graag op mijn beurt mevrouw Moenis willen bedanken en feliciteren. Nee, ναι, broeder, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Μούνη και να πω ότι όντω έχει κάνει πολύ καλή δουλειά με την γνωμοδότησή, με την γνωμοδότησή της. Επίσης ε, θα ήθελα και μία ε, ε, έτσι, διευκρίνηση, γιατί θα ήθελα να μου πει γιατί στην τροπολογία 5, στο δεύτερο τμήμα, προτείνει να διαγραφεί το τμήμα αυτό. Στο δεύτερο τμήμα, στην τροπολογία 5, γίνεται μία πρόταση ώστε στα πλαίσια της ε, ε, ΓΚΑΣΠ να υπάρξει μια ε, κατανομή, ανακατανομή. Νομίζω η κυρία Μονίσινο προτείνει να διαγραφεί. Δεν, δεν καταλαβαίνω γιατί. Θα ήθελα ίσως κάποια διευκρίνηση. Για ποιο λόγο το προτείνεται να διαγραφεί αυτό το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 5. Και επίσης να κάνω και ένα πιο γενικό σχόλιο. Το κοινοβούλιο αυτό και σε αυτή την γνωμοδότηση ζητά να εμπλακεί ε, άμεσα σε ό,τι αφορά και την προετοιμασία αλλά και τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση, τον έλεγχο των μέτρων που θα αναλυθούν. Και έναντι της ε, είπα της εκπροσώπου όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της, το είπαμε ότι θα πρέπει να μας συμπεριλάβει περισσότερο, να έρχεται να μας μιλά, να χρησιμοποιήσει το κοινοβούλιο ώστε να είμαστε και εμείς, αλλά και οι υπεύθυνοι βεβαίως των επικεφαλής των αντιπροσωπείων, να εμπλακούν περισσότερο στην όλη διαδικασία. Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε μια ακρόαση του εκπροσώπου για το Σουδάν. και στην ε, ακρόαση αυτή ούτε μία ούτε ε, δεν είδαμε πάνω από 7 ευρωβουλευτές. Ήταν λυπηρό ε, και παρόμοια πράγματα ζούμε κάθε, σχεδόν κάθε φορά. Ακόμη και όταν έγινε η ακρόαση με την υποεπιτροπή για την ασφάλεια και την άμυνα. Και εκεί λίγοι ήταν οι παριστάμενοι. Και πραγματικά ήταν ε, ντροπή να μην ε, παριστάμεθα όταν έχουμε τέτοια είδου ακροάσει. Θα ήθελα να καλέσω λοιπόν όλου. Εντάξει, μπορούμε όλοι να λέμε ε, ωραία λόγια και να ζητούμε να συμπεριλαμβάνεται το κοινοβούλιο περισσότερο στι όλε τι διαδικασίε, αλλά εν τω μεταξύ όμω πρέπει και το κοινοβούλιο να δείχνει την παρουσία του. Πρέπει να είμαστε ε, πολλοί όταν γίνονται τέτοιου είδου ακροάσει. Δεν μπορούμε να ζητούμε κάτι και μετά να μην είμαστε παρόντε ισχύει και για τη δική μου την ομάδα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ισχύει και για όλου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Νέης για το σχολείο σας το οποίο συμμερίζαμε. Το λόγο έχει η συγγεντρία για να απαντήσει. Αλλά εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δω αν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Όχι. Αν συμφωνεί λοιπόν η συγγέντρια, να ακούσουμε και την Κομισιόν. Παρακαλώ, ο κύριος Γκάρι Μίλλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδοκιμάζει την γνωμοδότηση της εισηγήτριας, γιατί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ξεκινήσει συζητήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εφαρμόσει το σκέλος ΚΕΠΑ της Διοργανικής Συμφωνίας ικανοποιώντα τι επιθυμίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βέβαια, δεν είναι μόνο συμβαλόμενο μέρο τη ε, Διοργανική Συμφωνία η Ευρωπαϊκή. Η Διοργανική Συμφωνία είναι τριμερή αυτή η συμφωνία και συνάπτεται μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε, στα πλαίσια των γενικότερων διαπραγματεύσεων μεταξύ των τριών συμβαλωμένων μερών θα πρέπει να συνεχιστούν οι διαβουλευσει. Έχουμε και το γραφείο του, της ΥΠΑ της εκπροσώπου και την, εξωτερική την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Η γνωμοδότηση αυτή θα συμβάλλει στη συζήτηση που θα ακολουθήσει με συμμετοχή όλων αυτών των ενδιαφερομένων. Σε ό,τι φορά την είπατε εκπρόσωπο, γνωρίζετε ότι προέβη σε μια εκτενή δήλωση για την ε, πολιτική λογοδεσία που έχει επισυναυθεί στην επίσημη κυβέρνηση και έχει επισυναυθεί και στην ε, ε, επίσημη απόφαση και στη δήλωση αυτή η κυρία Άστον ανέλαβε πολλές δεσμεύσεις για την ΚΕΠΑ. Μην ξεχνάτε τις παραγράφους 1, 8, και 10 της δήλωσης που αφορούν ιδιαίτερα αυτό το θέμα της ΚΕΠΑ, ότι εκπρόσωπος θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις συζητήσεις για τη διαμόρφωση της νέας διοργανικής συμφωνίας και έχει δεσμευθεί υπέρ της ενίσχυσης της διαφάνειας. Φυσικά οι λεπτομέρειες αυτής της διοργανικής συμφωνίας ε, θα αποτελέσουν αντικείμενο των μελλοντικών διαπραγματεύσεων. Σε ό,τι αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορούμε να σχολιάσουμε κάποιες τροπολογίες για τα δημοσιονομικά θέματα. Για παράδειγμα, την τροπολογία 5 που προτείνει τροποποίηση της διάρθρωσης του προϋπολογισμού. Βέβαια, αυτό είναι κάπως τεχνικό θέμα, αλλά οι δαπάνε στη ΚΕΠΑ περιορίζονται σε ένα κεφάλαιο του προπολογισμού, όπω προβλέπει η Διοργανική Συμφωνία. Υπάρχουν όμω ε, και υποδιαιρέσεις σε διάφορα άρθρα η τροπολογία σκοπεύει να διαγράψει όλη αυτή τη διάρθρωση των άρθρων, κάτι που δημιουργεί μια στάθεια στον προϋπολογισμό από χρόνο σε χρόνο. Οπότε θα πρέπει να αποφασίσουμε κάθε χρόνο τη δομή του προϋπολογισμού. Εμείς προτιμούμε μια σταθερή δομή προϋπολογισμού για λόγους διαφάνειας και λόγους ε, λογοδοσίας. Και στην ε, δημοσιονομική διαδικασία η Επιτροπή Προϋπολογισμών, όπως θα γνωρίζετε, τάχθηκε υπέρ της διασφάλισης της νέας ε, διάρθρωσης, αλλά και την δημιουργία νέων τριών δημοσιονομικών γραμμών για τις μεγαλύτερες αποστολές της ΚΕΠΑ, κάτι που θα βελτιώσει τη διαφάνεια, κάτι που ανταποκρίνεται στις ε, δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος στην δήλωσή της για την πολιτική λογοδοσία. Είπε ότι θα προσπαθήσει να βελτιώσει τη διαφάνεια για τις πιο σημαντικές ε, αποστολές της ΚΕΠΑ. Εμείς συμφωνούμε με την ε, τροποποίηση που έγινε στην Επιτροπή Προπολογισμών, αλλά αυτή η τροπολογία, η παριθμό 5, δεν συνάδει με τη γενική αυτή κατεύθυνση. Οι υπόλοιπε τροπολογίε για τα δημοσιονομικά είναι πιο τεχνικέ. Θα κοινοποιήσω τα σχόλιά μου απευθεία στην ε, εισηγήτρια. Με μερικέ ίσω υπάρχουν προβλήματα. Πάντω, από ό,τι ξέρω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επατή Εκπρόσωπο είναι υπέρ τη βελτίωση τη διαφάνεια και θα διαδραματίσουμε ενεργό ρόλο στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση της νέας διοργανική συμφωνία. Ευχαριστώ. Απάντηση λοιπόν και συμπέρασμα για την συγκήτρια. Σας ευχαριστώ. Κυρία Νέιτ, κατέθεσα την τροπολογία 5 για να μην περιορίσω τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου τις δημοσιονομικές ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Γιατί με την πρόταση δημιουργείται μια ανελαστικότητα. Άλλωστε το κεφάλαιο 4 του προϋπολογισμού είναι από τα κεφάλαια που περισσότερο υπάγονται στην ελαστικότητα για πρόβλεπτες καταστάσεις ή για σημαντικές αλλαγές στη δημοσιονομική πραγματικότητα. Και αυτό το κεφάλαιο είναι το μοναδικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού που χαρακτηρίζεται από τέτοια ακαμψία και σταθερότητα. Είναι το μοναδικό κεφάλαιο, το μοναδικό σταθερό κεφάλαιο του προϋπολογισμού, αν θέλετε. Γιατί στην Γεωργία, ας πούμε, δεν έχουμε συγκεκριμένη μνήμα του, της βρώμης, του ρυζιού, το, της μπανάνας. Γιατί να έχουμε τέτοια ακαμψία στην ε, δημοσιονομική πολιτική. Ήταν λογικό μέχρι στιγμής γιατί είχαμε απόλυτη οριοθέτηση των δαπανών, των κυβερνητικών δαπανών στις οποίες ε, δεν υπησερχόταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα όμως υπάρχει διεύρυνση αυτών των αρμοδιοτήτων, οπότε δεν έχουν νόημα αυτοί οι περιορισμοί και αυτή η ανελαστικότητα που χαρακτηρίζει τον προπολογισμό σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Νομίζω ότι έτσι αντίθετα ενισχύουμε τη διαφάνεια και την ε, συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις αποφάσεις. Βέβαια, όπως είπατε, η συμμετοχή θα πρέπει να είναι ενεργό συμμετοχή των Ευρωβουλευτών στις συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις συνεδριάσεις με την ύπατη εκπρόσωπο, αλλά χρειαζόμαστε και ένα θεωρητικό πλαίσιο που θα επιτρέπει αυτή την ελαστικότητα και αυτή την ενεργό συμμετοχή. Και αυτό είναι ο στόχος της τροπολογίας 5. Δεν θέλουμε να περικόψουμε αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αντίθετα, θέλουμε να βελτιώσουμε την ελαστικότητα στον τρόπο ανάμειξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. κυρία Λόχμπίλερ, λέει η συγγετρία, ε, θέλουμε να προσδιορίσουμε το πλαίσιο διαλόγου και με τα υπόλοιπα κοινοτικά θεσμικά όργανα σε θέματα προπολογισμού. Δεν προσδιορίζουμε το περιεχόμενο της ΚΕΠΑ. Στη γνωμοδότησή μου δεν υπησέρχομαι σε τέτοια θέματα ουσίας της ΚΕΠΑ. Αυτό γίνεται σε άλλε εκθέσεις και γνωμοδότηση. Και δεν είναι αντικείμενο της γνωμοδότησή μου το κατά πόσο οι αποστολές της ΚΕΠΑ θα έχουν στρατιωτικό χαρακτήρα ή όχι. Σε ό,τι αφορά τι συναντήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είμαι στη διάθεσή της για συνομιλίε προκειμένου να βελτιώσω τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχει άλλο. Περνάμε στο 6 το επιχείρημα του 6 είναι η δημιουργία μια ε, συγκρότηση μάλλον ενωσιακού μηχανισμού ταχεία αντίδραση. Αυτό ο μηχανισμό ταχεία αντίδραση τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σαφεί επιπτώσει σε επίπεδο εξωτερική πολιτική και άρα <coughs> πρέπει να τονιστεί η κοινοτική του πτυχή και γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε, συντάξουμε αυτή τη γνωμοδότηση για την Επιτροπή ε, Ανάπτυξης στην οποία έχει ανατεθεί η βασική αρμοδιότητα για αυτό το θέμα και Μα ζήτησε να συντάξουμε μια γνωμοδότηση επί τη βάση του άρθρου 50 του κανονισμού. Η συγκίτρια του είναι η κυρία Βέμπερ που είναι στην αίθουσα και στην οποία δίνω αμέσω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ε, αναφέρατε μόλις, Η έκθεση για την ταχεία αντίδραση στι κρίσει είναι μια έκθεση για την Επιτροπή Ανάπτυξη. Ε, συζητήθηκε, συζητήθηκε χθε το απόγευμα στην Επιτροπή Ανάπτυξη και η Επιτροπή ΑΦΕΤ αποφάσισε να δώσει μια γνωμοδότηση για την έκθεση αυτή. Θα πρέπει να αναφέρω ότι στην ΤΕΒΕ είναι μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας και ότι η Επιτροπή θα προβεί σε μια ανακοίνωση για τη δημιουργία της, του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης στα τέλη αυτού του χρόνου. Άρα λοιπόν η έκθεση της ΔΕΒΕ και, αυτής της επιτρο... και, αυτή η θα πρέπει να θεωρηθούν ως βήματα σε μια ευρύτερη όμως διαδικασία. Από την άποψη της ΑΦΕΤΟΜ τώρα, Στη γνωμοδότηση που εγώ συνέταξα ήθελα να τονίσω κάποια πράγματα που κατά την άποψή μου είναι πολύ ε, σημαντικά για την Επιτροπή μας. Νομίζω ότι το πρώτο βασικό βήμα στην προσέγγιση της ΑΦΕΤ είναι ο ρόλος ε, του Αντιπροέδρου, του, του του εκπροσώπου στην Κομισιόν στο συντονισμό όλων των κοινοτικών δράσεων σε τρίτες χώρες και περιφέρειες. Και ως προς αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι οι μέθοδοι εργασία και οι δομές που υπάρχουν για την ε, εξωτερική υπηρεσία με τις κατάλληλες αρμοδιότητες ε, για τους ε, εκπροσώπους μας εκεί ε, θα πρέπει να αναφέρονται στη γνωμοδότηση. Επίσης αναζητούμε την σαφήνεια και τη διαφάνεια καθώς και το συντονισμό με άλλα κοινοτικά μέσα όπως αυτό που υπάρχει υπό την CFTP, την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, αυτά δηλαδή που ήδη υπάρχουν ή που θα συσταθούν κατόπιν μιας καταστροφής. Είναι όντως πολύ σημαντικό να είμαστε αποτελεσματικοί. Είναι ζωτική σημασία όταν κανείς θέλει να ανταποκριθεί σε καταστάσεις κρίσης. Ακριβώς αυτό σημαίνει ταχύ αντίδραση, σημαίνει αποτελεσματικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις οικονομικέ ε, περιστάσεις τι οποίες βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ένωση, διότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας και που μπορούν να διαθέσουν η Ένωση και τα κράτη-μέλη σε τέτοιες περιπτώσεις. <clears throat> Τώρα, για την στρατιωτική πτυχή και πώς θα μπορούσαμε ή αν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε σε περιπτώσεις κρίσης. Η γνωμοδότηση αναφέρει ότι αυτή θα πρέπει να είναι η έσχατη λύση, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές του Όσλο όσον αφορά την, τα στρατικά μέσα και δυνατότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ε, ανακούφιση των πολιτών σε περιπτώσεις καταστροφής. Όμως θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι κάθε κρίση έχει τις ιδιαιτερότητές της και ανάλογα με την κατάσταση σε, κάποιες, σε κάθε χώρα και σε κάθε περιφέρεια οι στρατιωτικές ε, δυνατότητες μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο Τονίζουμε πλέον ότι ο ΙΕ θα πρέπει να παίξει συντονιστικό ρόλο και σίγουρα θα πρέπει να παραβληθεί στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας αντίδρασης ή ανταπόκρισης. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε για όλους τους διεθνείς φορείς που επιτόπου ασχολούνται με τη βοήθεια σε περιπτώσεις καταστροφών. Πρόεδρε, αναφέρατε κάτι όσον αφορά το αίτημα της ΑΦΕΤ να γίνει μια κοινή έκθεση με την Επιτροπή Ανάπτυξης. Λυπάμαι, αλλά δεν κατάλαβα ακριβώ ποια ήταν η απάντησή σας. Μήπως μπορείτε να επαναλάβετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Με ρωτήσατε και αφορά την από κοινού σύνταξη της έκθεσης με την ΤΕΒΕ επί τη βάση του άρθρου 50. Ναι, όντως περί αυτού πρόκειται. Ζητήσαμε να χρησιμοποιηθεί, να ισχύσει το 50 για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ε, από κοινού με την ΤΕΒΕ ακόμα και αν είναι σε διαφορετικούς ε, οδούς. Διαφορετικέ οδού. Ερώτημά μου είναι, έχουμε απάντηση σε αυτό το αίτημα. Όχι. Ακόμα δεν έχουμε απάντηση. Ίσως στο Στρασβούργο. Θα έχουμε άλλες παρεμβάσεις. Πρώτο, ο κύριος Γκάλερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομα να πω κάτι για το ΕΛΚ. Ο συνάδελφο Ντανζό είναι ο ε, σκιώδη ηγητή, δεν μπορούσε όμω να είναι παρόν σήμερα, οπότε εξ ονοματό του θα ήθελα και εγώ να κάνω ένα σχόλιο. Και θα περάσω στα αγγλικά. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Βέμπερ. Νομίζω ότι η γνωμοδότηση αυτή είναι όντω μια πολύ καλή βάση για να δουλέψουμε. Η έκθεση Ντεβί όντω ε, ε, επικεντρώνεται στην ε, πολιτική προστασία και στην ανθρωπιστική βοήθεια, οι οποίε είναι οι δύο βασικέ διαστάσει όταν μιλούμε για απάντηση σε τέτοιε περιπτώσει. Και εντάσσεται βέβαια και στα διαθέσιμα μέσα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να απαντά. Ε, σε τέτοιε περιπτώσεις. Πρέπει λοιπόν να έχουμε σωστό συντονισμό. Είναι ουσιώδου σημασία ο πρόεδρος και την πρόεδρος της Επιτροπής να μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο ώστε να εξασφαλίσουν μια καλή πολιτική και στρατιωτική συνεργασία και να υπάρχει μια συνολική προσέγγιση όταν θέλουμε να επέμβουμε έγκαιρα. Mm-hmm. Αυτή η πτυχή περιλαμβάνεται μέσα στην νομοδότηση αλλά θα θέλαμε να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Ε, η κυρία Άστον είναι αυτή που είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό τη συνολική απάντηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να έχει την κατάλληλη εντολή που θα της επιτρέπει να ενεργοποιεί αυτό το, αυτούς τους μηχανισμούς ανταπόκρισης στις ε, καταστροφές για να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσει να λειτουργεί άμεσα χωρίς να χρειάζεται την άδεια του Συμβουλίου κάθε φορά. Σε ό,τι αφορά τώρα το να χρησιμοποιήσουμε στρατιωτικά μέσα, όταν τα πολιτικά μέσα δεν είναι διαθέσιμα ή δεν είναι επαρκή, θα μπορούσαμε ίσως να βασιστούμε σε επιχειρήσεις της ΚΕΠΑ, όπου όπως αναφέρεται και στην νομοδότηση, ε, θα έχουμε ούτως ή άλλως και το Ταμείο Startup, το οποίο αναφέρεται και στην, ε, στο άρθρο 41 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε ο ύπατος θα έχει μεγαλύτερη δικαιοδοσία να αναλάβει δράση. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και άλλα στρατιωτικά εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν και να είναι χρήσιμα, όπως καλύτερες ομαδοποίησεις ή, ή α, ε, η μονάδα ε, αεροπορικών μεταφορών από το Αιτχόβεν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ε, εγώ θα συνεργαστώ και το ΕΛΚ με την συγκήτρια και θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες. Γενικώ, η έκθεση μιλά για την, η έκθεση μιλά για την, για την απάντηση σε καταστάσεις εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έπρεπε όμω να δούμε και το τι γίνεται εντός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, κυρίως ό,τι αφορά και την ρήτρα αλληλεγγύη που προκύπτει από την συνθήκη της Λισαβόνα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εκδρομοδότηση αυτή που κατευθύνεται προς τη σωστή κατεύθυνση Όσον αφορά την ουσία, όλοι συμφωνούμε στην ανάγκη να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη και πρακτική προσέγγιση ως ανταπόκριση στις καταστροφές. Καταρχήν θα πρέπει να αναπτυχθεί ο συντονισμός και η συνεργασία ανάμεσα στις πολιτικές και στις στρατιωτικές δυνατότητες και αυτό το θέμα είναι που συζητάμε σήμερα. Επίσης θα πρέπει να βελτιωθεί η προβλεψιμότητα και ως εκ τούτου η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης, ένα στοιχείο που επίσης περιλαμβάνεται στο κείμενο και τέλος ε, να ε, γίνουν σημαντικά βήματα για τη θέσπιση μιας ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολιτικής Προστασίας όπως αυτή που βλέπετε στην έκθεση Μπαρνιέ. Το στοιχείο αυτό λοιπόν συμπεριλαμβάνεται εδώ. Το στοιχείο που δεν συμπεριλαμβάνεται ωστόσο στη συζήτησή μας είναι η πρόβλεψη του άρθρου 214 παράγραφος 5 τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, που καλεί για τη δημιουργία ενός, ε, μιας ευρωπαϊκή θελοντικής, εθελοντικής δύναμης βοήθειας. Και θέλω να διαβάσω τη διάταξη τη συνθήκη, όπως σας είπα, είναι το άρθρο 214, παράγραφος 5 και λέει τα εξή. Με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου για κοινή συνεισφορά από νέους Ευρωπαίους στον ανθρωπιστικέ ε, δραστηριότητες βοήθειας της Ένωσης θα πρέπει να δημιουργηθεί, θα συσταθεί μια ευρωπαϊκή δύναμη ανθρωπιστική βοήθειας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο λειτουργώντας με την ε, συνήθεια νομοθετική διαδικασία θα ορίσει τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη λειτουργία αυτού του σώματο. Νομίζω κύριε Πρόεδρε και συνάδελφοι ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική διάταξη τη ε, συνθήκη που θα μπορούσε και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο κείμενο αυτό, το κείμενο που συζητάμε δηλαδή σήμερα. Θα πρέπει να δώσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες και κυρίως στους νέους μας ένα πλαίσιο ώστε να μπορούν ενεργά να συμμετέχουν σε προγράμματα που σχετίζονται με την ανθρωπιστική βοήθεια, την πολιτική προστασία και την ε, πήγουσα βοήθεια σε περίπτωση ε, προβλημάτων σε, σε περίπτωση ε, καταστροφών. Θα μπορούσαμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την, ε, την εμπειρία του ΟΗΕ και τέλος, για να κλείσω την παρέμβασή μου, να σας πω ότι πιστεύω πως όλα αυτά μπορούν να εξασφαλιστούν μέσω της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Εθελοντικού Σώματος Ανθρωπιστικής Βοήθειας όπως προβλέπεται από τη συνθήκη και είναι ένα στοιχείο πιστεύω πως αυτό πολύ εύκολα θα μπορούσε να ενσωματωθεί σε αυτό το κείμενο πράγμα που θα ήταν και σοφό κατά την απόψή μου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Επόμενη παρέμβαση η κυρία Λούζινγκ. Ευχαριστώ. Ως σκιώδης εισηγήτρια θα μιλήσω από την ΚΟΕ και να πω από την αρχή ότι την γνωμοδότηση έτσι όπως ε, έχει δεν μπορούμε να την δεχτούμε. Και εδώ βασικό σημείο κριτικής είναι η σύνδεση πολιτικών και στρατιωτικών εργαλείων που αναφέρονται και τονίζονται και ζητούνται μέσω της γνωμοδότησης. Επίσης, τον θετικό ρόλο της ε, ε, πολιτικής ε, δεν μπορούμε να τον δεχτούμε ακριβώς λόγω του ότι υπάρχουν αυτά τα, αυτά τα πετήματα, τις, αυτά αυτές οι απαιτήσει της σύνδεσης μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών επιχειρήσεων. Νομίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη, ε, ε, μεγάλο έλλειμμα δημοκρατίας στην ε, υπηρεσία εξωτερικών σχέσεων. Ε, τώρα, για την αντιμετώπιση των κρίσεων και τη χρήση των, στρατιωτικών δυνάμεων σε περίπτωση καταστροφών. Ακόμη και όταν μιλούμε για καταστροφές όπου τα πολιτικά εργαλεία δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους ή την υποδομή για να αντιμετωπίσουν παρκώς και πλήρως αυτές τις καταστροφές, αυτό είναι συνέπεια της ε, έλλειψης πολιτικής βούλησης. Δεν είναι νόμος της φύσης, δεν είναι ε, φυσική ε, απόρρια των πραγμάτων. Τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να έχουν την κατάλληλη χρηματοδότηση ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστροφές χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνουμε πάντα στη χρήση στρατιωτικών μέσων. Δεν μπορούμε πάντα να εξοπλίζουμε συνέχεια τα κράτη ώστε να, έχουμε, να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους καταστροφές μόνο στρατιωτικά. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι πεδίο διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλω τώρα να μπω σε άλλες λεπτομέρειες. Εμείς εμένουμε στο ότι οι καταστροφές δεν θα πρέπει να, να οδηγούν σε επέμβαση στρατιωτικών δυνάμεων. Και να κάνω και ένα σχόλιο που αναφέρεται στο, στη σημείο 3. Ακόμη και εάν ε, αρνηθούμε αυτό που προτείνεται. Αυτό που λέει το 3 θεωρώ ότι είναι ε, θετικό. Είναι θετικό να λέμε ότι τα στρατιωτικά μέσα είναι η τελευταία διέξοδος, η τελευταία λύση. Αλλά αυτό αντιτίθεται στο πνεύμα της νομοδότησης και στην γενική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί εκεί βασικός στόχος είναι να ενωθούν οι πολιτικές επιχειρήσεις με τις στρατιωτικές, ώστε να αποτελέσουν ένα κομμάτι της, ε, της ε, αντίδρασης σε τέτοιες καταστροφές. Κάτι λοιπόν που είναι θετικό, ε, οδηγείται ουσιαστικά, γίνεται κενό νοήματο σε άλλο σημείο, όπως αυτό που σας αναφέρω τώρα. Έχουμε δει ε, αποτελέσματα και στο Αφγανιστάν και σε άλλες χώρες. Είχαμε κάνει πολλές ακροασει, ε, ε, ακούσαμε πάρα πολλού οργανισμούς που παρεμβαίνουν και πάντα το θέμα ήταν ότι γίνεται και χωρίς την στρατιωτική παρέμβαση να λυθούν οι καταστάσει αυτέ και δεν χρειάζεται πάντα να παρεμβαίνει ο στρατό. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς, η Επιτροπή. Όχι. Α, ναι, ναι. ωραία. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ονομάζομαι Πίτερ Μπελίν. Είμαι υποδιευθυντής στην Γενική έκο στην Μονάδα για την Πολιτική Προστασία. Σας ευχαριστώ για την γνωμοδότηση και τις προτάσεις προ το Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ιδιαίτερα το ζωηρό ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ε, κρίσεων και καταστροφών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι σημαντικό θέμα και για του Ευρωπαίου πολίτε. Το βαρόμετρο δείχνει ότι 90% των πολιτών περιμένουν πιο ενεργοδράση τη Ένωση σε περίπτωση καταστροφών. Είχαμε πρόσφατα διάφορα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση και άμεση αντίδραση σε καταστροφές. Και μάλιστα είχαμε και χρηματοδότηση 7,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τη διετία 2008-2010. Έτσι θα μπορέσουμε να πειραματιστούμε σε διάφορες νέες προτάσεις ό,τι αφορά την ταχεία αντίδραση σε περίπτωση καταστροφής. Μάλιστα, είχαμε και το ψήφισμα του Φεβρουαρίου του 2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ΑΕΤ. Και μάλιστα και η γνωμοδότηση ενστερνίζεται την ίδια προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ταχεία αντίδραση. Το 2010 είχαμε πολλές καταστροφές στην Αιτή. Το Πακιστάν ήταν δύο από τα πιο συγκλονιστικά παραδείγματα που χρειάστηκε να ανταποκριθούμε άμεσα και φάνηκε η δυνατότητα της παγκόσμιας κοινότητας ε, και τα όρια της παγκόσμιας κοινότητας να αντιδράσουν τέτοιου είδους ε, μεγάλες καταστροφές. Είχαμε και την περίπτωση της έκρηξης του ηφαιστείου στην Ισλανδία, πλημμύρες σε πάρα πολλές χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και στη Ρωσία ε, πυρκαγιές άνευ προηγουμένου. Είχαμε ενεργοποίηση του μηχανισμού αυτού μόνο φέτος 20 φορές, κάτι που δημιουργεί πολλά και διάφορα θέματα. Εν ώψη της, ε, του αυξανόμενου αριθμού και της περιπλοκότητας των καταστροφών θα πρέπει να δώσουμε ε, μεγαλύτερη έμφαση στα μέτρα μείωσης ε, των κινδύνων. Και έχουμε εντατικοποιήσει τις προσπάθειες και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στρατηγική πρόληψη, αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας την προσπάθεια μείωσης του κινδύνου στα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας. Και η ΑΕΤ και άλλες περιπτώσεις μας έδειξαν ότι ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης αντεδρούσε γενικώ καλά, αλλά λόγω των διαρθρωτικών περιορισμών της, για παράδειγμα η εξάρτησή της από εθελούσια προσφορά των κρατών μελών, δημιουργεί προβλήματα και αυτό έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα, την συνοχή αλλά και την προβλεψιμότητα σε ό,τι αφορά τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους επόμενου μήνε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει προτάσει προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη μορφή μιας ανακοίνωση για τη δυνατότητα αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση καταστροφών. Εκεί θα προτείνουμε συγκροτημένο και αποδοτικό τρόπο για την αντιμετώπιση αυτών των ε, καταστάσεων. Βέβαια το θέμα ετοιμότητα και ανταπόκριση η διαχείριση τέτοιων καταστάσεων ε, εναπόκειται και στι ε, κυβερνήσει, αλλά μια σωστή συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία. Βέβαια, όπως σας είπα, εξαρτώμαστε από ad hoc προσφορές και οικειοθελή ανάμειξη των κρατών μελών. Βέβαια, υπάρχει αναπόφευκτο και ένας βαθμός αυτοσχεδιασμού σε τέτοιες περιπτώσεις και οι αποφάσεις δυστυχώς δεν λαμβάνονται τόσο γρήγορα όσο θα επιθυμούσαμε. Πάντως, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα σύστημα που θα εξασφαλίζει σημαντικούς πόρους για άμεση δράση. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δοκιμάσει διάφορα σενάρια για σημαντικές καταστροφές. Επίσης θα δει τι δυνατότητες προσφοράς έχουν τα κράτη-μέλη για τέτοιου είδους άμεση δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ζητήσει από τα κράτη-μέλη να έχουν διαθέσιμες κάποιους πόρους σε περίπτωση που θα ανακύψουν καταστροφές προκειμένου να κινητοποιούνται άμεσα. Επίσης θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε κάποιες ρυθμίσεις ε, άμεσης μεταφοράς αυτής της ε, ανάπτυξης βοήθειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις τρίτες χώρες θα εξασφαλίσουμε καλύτερο συντονισμό των επιτελείων παρόλο που μερικές φορές ε, ο έλεγχος γίνεται από άλλους έξω κοινοτικούς παράγοντες. Σε Εξαιρετικέ περιπτώσει και σε έσχατη λύση μετά τι κατευθυντήριες γραμμές του Όσλο η πολιτική προστασία και η ανθρωπιστική ενίσχυση μπορούν να συμπληρωθούν και από στρατιωτικά μέσα. Για παράδειγμα ο στρατό μπορεί να ε, εξασφαλίσει τη μεταφορά. Θέλουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο να χρησιμοποιήσουμε κάποια στρατιωτικά μέσα και σε άλλες μορφές ενίσχυσης και προσπαθούμε να ευθύσουμε μια στρατηγική προσέγγιση και στα θέματα επικοινωνία. Πολλές φορές η αντίδρασή μας σε θέματα καταστροφών ήταν αποτελεσματική, αλλά δεν είναι αρκετά ορατή και αναγνωρίσιμη πάντα. Βέβαια η προβολή αυτή της ε, ανάμειξης δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά και το, κοινό, το ευρύ κοινό δικαιούται να γνωρίζει πώς παρέχει τη βοηθειά της Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια η ανακοίνωση είναι μόνο το πρώτο βήμα. Του χρόνου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει και νομοθετικές προτάσεις για την εφαρμογή των συστάσεων που θα περιλαμβάνει η επόμενη ανακοίνωση. Πάντως προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την κατάρτιση αυτής της νομοθεσίας και ελπίζω να μας υποστηρίξετε ε, σε αυτές τις νομοθετικές προτάσεις που θα δώσουν σάρκα και οστά σε αυτές τις φιλόδοξες ιδέες. Σας ευχαριστώ. Η εισηγήτρια θέλει να ολοκληρώσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν στη συζήτηση και βεβαίως περιμένω να δω και τις τροπολογίες που θα υποβληθούν. Τώρα, σε ό,τι αφορά την χρήση των ε, στρατιωτικών ε, δυνάμεων χωρίς, ε, ως τελευταία λύση, χωρίς βέβαια να θέλω να μπούμε σε ιδεολογική συζήτηση, θεωρώ ότι είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες που έχει στη διάθεσή της. Οπότε όταν μιλούμε για στρατιωτικές υποδομές δεν ε, σκεφτόμαστε να ξεκινήσουμε τώρα πολέμους σε οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου, αλλά προσπαθούμε να, την, ε, να δούμε την επέμβαση της στρατιωτική ως ε, τρόπο για να λυθεί το πρόβλημα που έχει προκύψει. Βεβαίως οι συνάδελφοι είναι ελεύθεροι να υποβάλουν τις τροπολογίες τους για να διαγράψουμε κάποιες από τις ε, παραγράφους που αναφέρονται στη στρατιωτική παρέμβαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Κομισιόν για την παρέμβασή της. Μας δίνει έτσι και αυτή μια γεύση για το τι θα περιλαμβάνει η ανακοίνωση που θα μας αποσταλεί στις αρχές του επόμενου έτους και νομίζω ότι ως προς αυτό είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το δικό μας αίτημα να γίνει η ΑΦΕΤ συνεισηγητής για το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό, έχοντας υπόψη βεβαίως και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ε, συνάδελφε Βέμπερ. Να θυμίσω ότι η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι 7 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι. 26-27 Οκτωβρίου θα, συζητηθεί, ή θα ψηφιστεί έκθεση στην ε, Επιτροπή. Επόμενο θέμα έχουμε την χορήγηση εγγύησης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις για σχέδια εκτός της Ένωσης. Είναι γνωμοδότηση του κυρίου Πεγιόν Πολύ σημαντικό θέμα, που ανανεώνει ένα θέμα. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο, στο οποίο αποφασίζουμε με συναπόφαση με, και έχουμε και μια γνωμοδότηση της Επιτροπής των Σοφών μετά ε, ε, όσον αφορά τις ε, δραστηριότητες εκτός Ένωσης της ΕΤΕΠ. Μεγάλο το ενδιαφέρον όσον αφορά την ε, ΕΤΕΠ και το ρόλο της στη χρηματοδότηση της εξωτερικών δράσεων και κυρίως την χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας νέος ε, θεσμικός οργανισμός, είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, που αποτελεί και έναν απαραίτητο πλέον συνομιλητή για την ΕΤΕΠ. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Πέγιον για να μας κάνει την εισήγησή του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είπατε ήδη τα πιο σημαντικά πράγματα. Είναι αλήθεια ότι είναι σημαντικό για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να παίξει το πλήρη ρόλο της προς την Επιτροπή προπολογισμών, που είναι αρμόδια επί τη ουσία, διότι η ΕΤΕΠ στην εξωτερική της εντολή, την οποία αναθεωρούμε εδώ για δύο χρόνια, είναι το οικονομικό χέρι της ε, εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι το μόνο, αλλά είναι ένα από αυτά που μπορούν να δώσουν χρήματα. Δεύτερον, να το είπατε κι εσείς, ότι είμαστε εδώ σε διαδικασία συναπόφασης μετά από μια αναπόφαση την οποία ε, εφεσιβάλαμε ε, το Συμβούλιο. Άρα λοιπόν μπορεί να παίξει ρόλο το Ευρωπαϊκό, Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με την Επιτροπή Προπολογισμών και την Επιτροπή Ανάπτυξης ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ε, μια στεναρή άποψη. Έπειτα, μέσα στην ίδια τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με νέα στοιχεία Ναι, δεδομένα. Έχει ξεκινήσει ένας προβληματισμός, αναφερθήκατε στην έκθεση της Επιτροπής των Σοφών, της οποίας προέδρεψε ο κύριος Κοντουσούμ. όσον αφορά τα μέσα, τα χρηματοδοτικά που θα, έχουμε, ε, που θα έχει η τράπεζα, άρα και εμείς, για να ασκήσουμε την εξωτερική μας πολιτική τα επόμενα χρόνια. Πολύ σύντομα λοιπόν, εγώ προτείνω για να ανοίξει η συζήτηση, καταρχήν η Κομισιόν μάλλον το συνοψίσω γιατί το γνωρίζουν όλοι, μέσα στην πρότασή της ε, βάλει πέντε πολύ σημαντικές προ... προτάσεις. Μία προαιρετική εντολή που είναι μία προέκταση 2 δις ευρώ για τα προγράμματα που αφιερώνονται στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Ε, δεύτερον, που είναι κάτι που είναι πολύ διαφορετικό, και είναι μια αλλαγή στον τρόπο εργασίας της ΕΤΕΠ ότι δεν ορίζονται δηλαδή με περιφερειακό τρόπο οι στόχοι αλλά ε, ορίζονται οριζόντιοι στόχοι για πολιτικές οι οποίες δεν θα είναι στοχευμένες γεωγραφικά με τρεις βασικές πολιτικές, ε, ε, κλιματικές αλλαγές, ανάπτυξη οικονομικής και κοινωνικής υποδομής και ανάπτυξη του, ιδιωτικού τομέα, του τοπικού ιδιωτικού τομέα και κυρίως του μικρομεσαίες. Και εδώ υπάρχει και ένας ε, ένας οριζόντιος στόχος, δηλαδή η στήριξη τη περιφερειακή ε, ολοκλήρωση. Τρίτο θέμα είναι ο συντονισμό ανάμεσα στις πολιτικές τη ΕΤΕΠ και τις εξωτερικές πολιτικές τη Ένωσης. Θα πρέπει αυτά πάντοτε να προσαρμόζονται και κυρίως να ενισχυθεί η δυνατότητα της ΕΤΕΠ να στηρίξει του αναπτυξιακού στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, ε, πέμπτη πρόταση της Κομισιόν είναι η άμεση προέκταση της εντολής του ΙΣΕΤΕΠ σε πέντε νέες χώρες, Ισλανδία, Λευκορωσία, Λιβύη, Ιράκ και Καμπότζη. Εγώ προτείνω και φαντάζομαι θα είναι άποψη και των άλλων επιτροπών να στηρίξουμε μια συζήτηση για αυτές τις νέες χώρες αλλά και να στηρίξουμε τις τροποποίησεις της εντολής που προτείνει η Κομισιόν. Αυτό Ωστόσο θα πρέπει να μας προβληματίσει και περισσότερο και να προετοιμάσουμε τη συνέχεια, διότι διαβλέπουμε ποιε θα είναι οι προκλήσεις με τις νέες χρηματο... δημοσιονομικές προοπτικές και την επόμενη εντολή. Καταρχήν, ε, πρώτο ζήτημα, εάν θέλουμε η ΕΤΕΠ και άρα οι πολιτικές μας να παίξουν πλήρως το ρόλο τους, προτείνουμε να ενισχυθεί το μέσο αυτό με μια ουσιαστική αύξηση των ανώτατων ορίων χρηματοδότησης, και ιδιαίτερα επειδή πολλά χρήματα έχουν ήδη καταναλωθεί, αφού εισάγονται πέντε νέες χώρες τώρα, δηλαδή 2011-2013, αντίστοιχα με αυτή την γεωγραφική προέκταση να αυξηθεί η οροφή χρηματοδότησης που δίνεται επί τη βάση της εγγύησης της Ένωσης. Ταυτόχρονα επιθυμούμε η ΕΤΕΠ να αυξήσει τις δραστηριότητές της, αλλά ε, βασιζόμενοι περισσότερο στους ίδιους τις κινδύνους, διότι δεν χρειάζεται εγγύηση της Ένωσης για κάποια προγράμματα που δεν ανταποκρίνονται στους στόχους πολιτικής της Ένωσης. Άρα λοιπόν να γίνεται μεγαλύτερη διάκριση ανάμεσα στα προγράμματα τα οποία χρειάζονται αυτήν την κίνηση και αυτά που δεν τα χρειάζονται. Επίσης προτείναμε κάτι που δεν υπάρχει, και το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως εδώ και στην Επιτροπή ανάπτυξη την δραστηριοποίηση μιας εντολής 200 εκατομμυρίων ευρώ που θα είναι αφιερωμένα για τις μικρο... στις μικροπιστώσεις τέλος, αν χρειαστεί τελικά αύξηση των οροφών, αν υπάρξει και, και μεγαλύτερη και αποκέντρωση των δράσεων να αλλάξουν και οι μέθοδοι της ΕΤΕΠ ώστε να μπορούμε καλύτερα να αξιολογήσουμε και να παρακολουθήσουμε τα σχέδια καθώς και να έχουμε καλύτερες εκθέσεις για αυτά τα προγράμματα ώστε να αξιολογούμε την εργασία που γίνεται στην πράξη με μεγαλύτερη διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών. Αυτό θα γίνει γιατί, αυτό θα σημάνει βέβαια γιατί η ΕΤΕΠ αυτή τη στιγμή δεν έχει τη διάθεση της τα μέσα ούτε τα ανθρώπινα μέσα ε, τους ανθρώπινους πόρους, ώστε αυτοί να αφιερωθούν στις αναπτυξιακές δραστηριότητες της ΕΤΕΠ. Και επίσης έχουμε εισάγει συστηματικά, γιατί έχουν ασκηθεί διάφορες επικρίσεις, ε, διάφορα συστήματα λοιπόν προειδοποίησης και ενημέρωση ε, των ΜΚΟ και τη κοινωνία των πολιτών. Ταυτόχρονα αυτό αντιστοιχεί στου προσανατολισμού τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Να προσέξουμε ώστε η ΕΤΕΠ να μην χρησιμοποιεί οδού, ε, διάβλου πιστοτικού που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, για να το πω έτσι εφημιστικά, στην φοροδιαφυγή. Να, μπορούν, λοιπόν, να μπορεί λοιπόν να συνεργάζεται με τις άλλες, τους οργανισμού οργανισμούς σε αυτό το τομέα. Σε επίπεδο θεσμικό λοιπόν η ΑΦΕΤ θα πρέπει να είναι παρούσα στη συζήτηση που ανοίγει. Εξορθολογισμός των ε, χρηματοπιστωτικών μέσων με προσέγγιση είδατε ότι διάφορες εγκεκριμένε προσωπικότητες εκφράστηκαν υπέρ της, ε, της ε, συνεργασίας ανάμεσα στην ΕΤΕΠ και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Αντασυγκρότηση και την Ανοικοδόμηση, που, την ΠΕΡΔ που αυτή τη στιγμή είναι κάπως ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Έπειτα θα πρέπει να γίνει εξορθολογισμός των μέσων υπέρ της ανάπτυξης και άρα δημιουργία μιας πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναπτυξιακή συνεργασία. Είναι μια πρόταση που μπορεί να έχει νόημα από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διατηρήσει τη δυνατότητα να χειρίζεται και να ελέγχει τα όσα συμβαίνουν, πράγμα που συμβαίνει σήμερα γιατί οφείλει να εγγυηθεί τις ε, πολιτικές της Ένωσης. Κάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό και που έχει διαγκριθεί στο πλαίσιο διαφόρων άλλων εκθέσεων της Επιτροπής μας είναι βέβαια η περιφερειοποίηση των δραστηριοτήτων της ΕΤΕΠ. Ας πούμε, την θυμηθείτε την Ευρωμεσογειακή Τράπεζα που συζητήσαμε στην έκθεση για τη Μεσόγειο θα ρίχνουμε αυτή την εξέλιξη γιατί έτσι είναι κανείς πιο κοντά επί τόπου, να μπορεί πιο εύκολα να βρει εταίρους ε, τοπικούς αλλά φυσικά πάντα με τον έλεγχο από πλευράς της ε, ΕΤΕΠ αυτών των μέσων γιατί υπάρχουν ανησυχίες. Έπειτα, που το είπατε και εσείς Πρόεδρε, υπάρχει Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων και εδώ που επιμείναμε πολύ στις προτάσεις μας, ώστε το σύνολο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και ιδιαίτερα η εξωτερική υπηρεσία να εμπλακούν μέσα σε αυτή τη συνεργασία ανάμεσα στην Κομισιόν και στην ΠΕΗ το κοινοβούλιο όμως παίζει το ρόλο ότι υπάρχουν πολλές τροπολογίες λοιπόν που θυμίζουν αυτό που είχε κάπως ξεχαστεί, ότι δηλαδή πρέπει να ε, βρει το χώρο της και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για αυτή την πολύ σαφή σας ε, εισήγηση. Και τώρα το λόγο έχουν οι σκιώδεις εισηγητές. Η κυρία Γιαννάκου η πρώτη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, πράγματι η έκθεση αυτή αλλά ιδίω η γνωμοδότηση από την Επιτροπή μας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρώτον διότι σηματοδοτεί την εμπλοκή της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ευθέως δηλαδή την εξωτερική πολιτική της Ένωσης στα ζητήματα που έχουν σχέση με την ανάπτυξη άρα και τα συμφέροντα της Ένωσης ε, και δεύτερον διότι μέσω της έκθεσης των σοφών που μας έχει παραδοθεί κατά κάποιο τρόπο διακρίνουμε αν μέχρι σήμερα η πολιτική αυτή έχει υπάρξει επιτυχής, δηλαδή η χορήγηση δανείων και εγγύσεων σε ε, τρίτες χώρες εκτός Ένωσης. Αν θέλει να μιλήσει κανείς περισσότερο επί της ουσίας, βέβαια θα αναρωτηθεί αν ταυτίζονται πάντοτε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα με τους στόχους ανάπτυξης των τρίτων χωρών. Πρέπει να ομολογήσουμε πως αυτό δεν είναι βέβαιο. Αν δηλαδή αυτό που θεωρείται ευρωπαϊκό συμφέρον ταυτόχρονα αποδίδει αναπτυξιακά στις τρίτες χώρες. Δεύτερον, ένα ερώτημα που θα πρέπει να θέσουμε στους αυτούς μας είναι ε, ποια είναι η πραγματική επιτυχία σε σχέση με τους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής γενικότερα παρακολουθώντας τα πράγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 80 ακόμα, εγώ προσωπικά θα σας έλεγα πως ούτε σαφείς απολύτως εκθέσεις υπάρχουν, ούτε είναι βέβαιο ότι η αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης έχει πετύχει ως αναπτυξιακή πολιτική. Πιθανόν να έχει ε, ενισχύσει τα συμφέροντα ε, οικονομικών παραγόντων της Ένωσης, εταιριών κτλ. Αυτό είναι βέβαιο αλλά ότι ε, έχει πετύχει σε σχέση με τους στόχους, αυτό είναι αμφίβολο. Βέβαια αυτό θα το εξετάσει η Επιτροπή Ανάπτυξης, ε, κύριε Πρόεδρε. Ο συνάδελφός μας κύριος Πεγιών, έχει κάνει μια σωστή κατά τη γνώμη μου αιτιολογική έκθεση και στηρίζει επίσης τις, ε, τα 500 εκατομμύρια των μικροπιστώσεων που πρέπει να δοθούν για μικρότερα έργα ε, αυτό που εγώ ήθελα να επισημάνω είναι ότι πριν από πολλά χρόνια είχαμε επενδύσει πάρα πολλά σε, στις τοπικές οργανώσεις στις τρίτες χώρες, δηλαδή σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, ε, σε μικρά ιδρύματα οικονομικού χαρακτήρα κλπ. Εγώ θέλω να εκφράσω έτσι πολλές αμφιβολίες αν αυτές οι οργανώσεις σε τοπικό επίπεδο υπήρξαν επιτυχείς ή αν έγινε σωστή δουλειά σε αυτό το επίπεδο. Ωστόσο δεν μπορούμε να αρνηθούμε να υπάρξουν ε, κάποια μικρά έργα που ίσως είναι αναγκαία και μπορούν να βοηθήσουν επιτόπου να καταπολεμηθεί ε, η απόλυτη φτώχεια που υπάρχει σε ορισμένες χώρες. Ε, είμαστε θετικοί για την έκθεση του συναδέλφου. Απλά θα ήθελα να σημειωθεί ίσως, αν ήθελε ο κύριος Πεγιών μέσα στην αιτιολογική έκθεση, ε, κατά κάποιο τρόπο να σημειωθούν τα ερωτηματικά που προκύπτουν ε, για όσα ανέφερα προηγουμένως ε, και κυρίως να δοθεί έμφαση στο ζήτημα που έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και πώς πρέπει και μπορεί να συνεργάζεται με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και άρα κατά κάποιο τρόπο να υπάρχει ένα είδος ελέγχου και από τη δική μας Επιτροπή, όχι μόνο από την ε, ε, Επιτροπή Ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Γεννάκου. Επόμενος είναι η σκιώδη συζήτρια Χάουταλα. Thank you very much, Chair. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το θέμα της ε, έκτασης αυτής της χρηματοδότησης ε, της ΕΤΕ που πέρυσι ήταν ε, σημαντικότερο και από τις παγκόσμιες τράπεζες και ουσιαστικά η, η γεωγραφική εμβέλεια της ΕΤΕΠ καλύπτει όλο τον κόσμο οπότε θα πρέπει να βελτιώσουμε τη, τη συνοχή και τη συνεκτικότητα αυτού του θεσμικού οργάνου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και πώς θα προσαρμόσουμε στους συνολικούς στόχους της ΚΕΠΑ. Συμφωνώ ότι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους είναι να αυξήσουμε τη συμμετοχή ε, του θεσμικού αυτού οργάνου σε θέματα ανάπτυξης και η ανάπτυξη είναι υπερισχύει της οικονομικής αποδοτικότητας ή της κερδοφορίας των σχεδίων. Και ευχαριστώ την Επιτροπή που πρότεινε καταμέτρηση του αντικτύπου των ε, σχεδίων, η εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδίων πριν τη χρηματοδότησή τους. Πριν πάντως ε, ε, προβούμε σε αύξηση της χρηματοδότησης της ΕΤΕΠ, θα πρέπει να εξετάσουμε πρώτα απ' όλα τους μηχανισμούς και κατά πόσο συνάδει η χρηματοδότηση της ΕΤΕΠ με τους ε, αναπτυξιακούς και άλλους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε την διαφάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και μάλιστα την περασμένη εβδομάδα είχα συζήτηση με τον κύριο Κιφόρο Διαμαντούρο, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τον ρώτησα πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενισχύσουν τα δικαιώματα, το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών, των Ευρωπαίων πολιτών για το τι συμβαίνει σε τρίτες χώρες. Γιατί αυτή είναι διαφάνεια. Και μου είπε ο κ. Διαμαντούρος ότι κάθε φορά που συνομιλεί με εκπροσώπους της ε, ΕΤΕΠ επιμένει στην ανάγκη ενημέρωση των πολιτών για τα σχέδια μεγάλης κλίμακας τουλάχιστον που χρηματοδοτεί η ΕΤΕΠ. Και χαίρομαι που και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά ιδιαίτερα η Επιτροπή μα, υποστηρίζει την προσέγγιση και το βασικό αυτό στόχο που έχει ο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, την αύξηση τη διαφάνεια, δηλαδή και τη ενημέρωση του κοινού. Μερικά ε, σχέδια και προγράμματα ευρεία κλίμακο έχουν και σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Και αυτό είναι το σημαντικότερο μέχρι, ήταν το σημαντικότερο μέχρι στιγμή ε, σκέλο τη μελέτη επιπτώσεων. Αλλά υπάρχει και το θέμα της επίπτωσης σε τοπικές και περιφερειακές συγκρούσεις. Και, αυτή, και αυτός ο αντίκτυπος θα πρέπει να εκτιμηθεί πριν ληφθεί η απόφαση χρηματοδότησης. Και πριν την απόφαση για την αύξηση της χρηματοδότησης, ελπίζω ο εισηγητής να τονίσει την ανάγκη συνοχής με τους ε, ευρωπαϊκούς ε, στόχους πολιτικής. Ιδιαίτερα στην εξωτερική πολιτική θα πρέπει να εξετάσουμε αν θα συμφωνήσουμε με την συμπερίληψη της Λευκορωσίας στις χώρες αποδέκτες. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει καν μία χειρονομία εκ μέρους της Λευκορωσίας ό,τι αφορά τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του εκδημοκρατισμού αυτής της χώρας. Το θέμα αυτό παραμένει εκρεμές. Ακόμη και η πρόταση για τα και τις μικροπιστώσεις, τα 500 εκατομμύρια. Καταπληκτική ιδέα, αλλά μπορούμε να βελτιώσουμε τους υπόλοιπους μηχανισμούς ώστε όντως ε, η χρήση αυτών των 500 ε, εκατομμυρίων να είναι βιώσιμη και να, ε, εξυπηρετήσει την υλοποίηση των στόχων που μας ενδιαφέρουν. Ευχαριστώ κύριο Χουντής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και η γνώμη της ομάδας μας είναι ότι ο κύριος συνάδελφος έχει κάνει μια πολύ σοβαρή και συστηματική προσπάθεια με τη γνωμοδότηση και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Όμως θα ήθελα κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι να σας πω ότι την ομάδα μας σε σχέση με τη γνωμοδότηση και το θέμα που συζητάμε το σοβαρό την απασχολούν τρία θέματα. Το πρώτο, η σύνδεση και η αναφορά και στο κείμενο και στην προφορική παρουσίαση αλλά και από όλους τους ομιλητές της δραστηριότητας και της χρηματοδότησης που δίνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με την εξωτερική πολιτική και τους πολιτικούς στόχους της Ένωσης είναι ένα ζήτημα πολύ συζητήσιμο, ήδη αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι. Η δική μας άποψη, όπως θα γνωρίζετε, την επαναλαμβάνω, έχουμε πολλές επιφυλάξεις, είμαστε αρνητικοί σχετικά με την πραγματική κατεύθυνση φιλιρινική και βοήθειας των αδύνατων χωρών από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι αυτή η πολιτική πάντα. Τις περισσότερες φορές μάλλον είναι στην αντίθετη κατεύθυνση. Επομένως, αυτό το στοιχείο, αυτό το πλαίσιο, αυτά τα κριτήρια σχετικά με το πλαίσιο δράση της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ε, μας κάνει πολύ ανήσυχους. Είμαστε επιφυλακτικοί ενδεχομένως να καταθέσουμε και τροπολογίες στα σχετικά σημεία προκειμένου να τοποθετηθεί κατά τη γνώμη μας καλύτερα το θέμα. Επιτρέψτε μου λίγο παραπάνω ανάλυση. Ε, αναφέρθηκε και πριν ...η στόχοι, οι εξωτερικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ανάπτυξη των χωρών στο οποίο δίδεται βοήθεια δεν είναι πάντα συμβατή. Θα έλεγα αν, και αυτή είναι η δική μας άποψη, οι προσπάθειες και η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προσβλέπει κυρίως στην ανάπτυξη, στην αντιμετώπιση κοινωνικών περιβαλλοντικών ζητημάτων είναι σίγουρο, μακροχρόνια ενδεχομένω, ότι αποφορτίζει το διεθνέ σκηνικό από αιτίε ένταση που δημιουργούνται από αυτά τα προβλήματα. Και επομένω είναι σε μια σωστή, κατά τη γνώμη μου, φιλιρινική, κατά τη γνώμη μας, φιλιρινική κατεύθυνση. Το δεύτερο σημείο που μα ανησυχεί, σφόδρα θα έλεγε κανεί, είναι η έμεση, μάλλον άμεση σύνδεση τη ε, δράσης της Ευρωπαϊκής Επενδύσεων με την νεοσύστατη υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Αυτό αναφέρεται σε αρκετά σημεία. Ο συγητής προτείνει να συμμετέχει η Επιτροπή, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στις προπαρασκευαστικές εργασίες σχετικά με τις πράξεις. Στην τροπολογία 10 αναφέρομαι. Όπως ξέρετε κύριε συνάδελφοι και κύριε Πρόεδρε, η ομάδα μας είναι ιδιαίτερα επιφυλακτική για το ρόλο και τις κατευθύνσεις αυτού του οργάνου. Και πολύ περισσότερο κυρίως που είναι καθαρό πια ότι έχουμε μια εμπλοκή πολιτικών και στρατιωτικών μέσων, με το οποίο προφανώς δεν συμφωνούμε. Άρα η εμπλοκή αυτής της νεοσύστατης, αμφισβητούμενης κατά μία έννοια, αμφιλεγόμενης γενικώ υπηρεσίας, μας α, δημιουργεί πολλές ανησυχίες και δεν συμφωνούμε με αυτή την σύνδεση. Και το τρίτο, επί της αρχής, ε, ότι νομίζω ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε γενικώ από την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεγαλύτερη συμμετοχή, όχι μόνο ενημέρωση όπως αναφέρεται εκεί από την Επιτροπή και πληροφορίες, αλλά αν είναι δυνατόν και στο επίπεδο του σχεδιασμού. Ταυτόχρονα θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζουμε ορισμένες από τις τροπολογίες του συναδέλφου που είναι σε θετική κατεύθυνση, όπως είναι η αύξηση των ανωτάτων ορίων χρηματοδότησης, η ενίσχυση των μικροπιστώσεων και βεβαίως θέλω να υπογραμμίσω το γεγονός και το στηρίζουμε ότι στο πεδίο εφαρμογή της εγγύησης αποκλείει κάθε δραστηριότητα που με άμεσο ή με έμεσο τρόπο σχετίζεται με οποιαδήποτε μορφή φοροδιαφυγής. Είναι θετικό αυτό και μακάρι να πραγματοποιηθεί. Κάθε μορφή φοροδιαφυγής ή χρήση χρηματοπιστωτικών ε, σχημάτων που βρίσκονται σε υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα και άλλες μορφές φοροδιαφυγής offshore εταιρείε. Αυτό το υποστηρίζουμε. Τελειώνοντας, ε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι η ομάδα μας είναι επιφυλακτική θα καταθέσει τροπολογίες στα ζητήματα που σας ανέφερα και τα οποία τα θεωρούμε σημαντικότατα και επίσης στο σημείο που πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο να χρηματοδοτούνται ε, έργα αποτροπής αν θέλετε της κλιματικής αλλαγής και όχι μόνο προσαρμογής αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε. Το λόγο ο κύριος Αλαβράκος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, προσωπικά πιστεύω ότι η οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο βεβαίω επιβάλλει τη διεύρυνση του τραπεζικού δανεισμού. Πιστεύω συνάμα ότι ένα τραπεζικό δανεισμό, εάν δεν είναι επαρκή για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης ή των χρηματοδομένων σκοπών, στην ουσία δεν είναι οικονομικός δανεισμός. Ε, δεν έχει καμία σημασία και δεν παράγει κανένα οικονομικό αποτελέσμα. Φοβάμαι λοιπόν ότι παρότι συμφωνώ στο σχέδιο της γνωμοδότησης και στο σχέδιο της συνοπτικής αιτιολόγησης του συναδέλφου του κ. Πέιλον και για την αύξηση του ποσού των 500 εκατομμυρίων και των 200 αντίστοιχα, είναι ποσά τέτοια τα οποία δεν καλύπτουν ανάγκες των λαών ή των χωρών στις οποίες ε, θα χορηγηθούν αυτά τα χρήματα υπό την εγγύηση βεβαίω της Ευρωπαϊκής Ένωση, που θα κάνουν τόσο αισθητή την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τα εντεύθυνα αποτελέσματα, δηλαδή την αναγνώριση και την ε, ε, σύναψη σχέσεων τέτοιων οι οποίες θα μας βοηθήσουν να έχουμε διεύρυνση της επιρροής μας στις τρίτες αυτές χώρες όσο και ως προς το αποτέλεσμα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φοβάμαι ότι θα χαθούν πολλά από τα χρήματα αυτά χωρίς να φέρουν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τι θα έλεγα. Θα έλεγα ότι όταν διψάει η αυλή μας και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπετε ότι έχουμε τεράστια προβλήματα και στην Ιταλία και στη Γαλλία και στην Ισπανία και στο Βέλγιο εδώ και στην Ελλάδα αλλά και στη Γερμανία από την ανάποδη πλευρά εκεί ζητούν λεφτά παραπάνω, εκεί ζητούν αυξήσεις, ενώ ε, ε όλες οι άλλες χώρες ζητούν τη μείωση των μειώσεων. Ε, πιστεύω ότι ίσως δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος να δώσουμε αυτά τα λεφτά. Να τα, στην ουσία να τα σπαταλήσουμε αυτά τα λεφτά σε τρίτες χώρες χωρίς κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Δεν θα παράξουμε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Πιστεύω λοιπόν ότι ίσως θα πρέπει να μελετήσουμε το θέμα πώς θα διευρύνουμε την συμμετοχή στον τραπεζικό δανεισμό των μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων που πλήττουν από την κρίση στην μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την ΕΤΕΠ, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να είμαστε πολύ περιορισμένοι στις διευρύνσεις μας σε τρίτες χώρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Πριν δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και της ΕΤΕΠ και μετά στον ε, εισηγητή Πεγιόν, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η διορία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 7η Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι. Αν δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο, να δώσω το λόγο στον κύριο Κιαρούν Καζόνη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Πεγιόν για την ε, εύστοχη έκθεσή του που περιλαμβάνει και πολλές καινοτόμες ιδέες, ακόμη και σε σχέση με τη δική μας ε, πρόταση και να ευχαριστήσω εκτός από τον κύριο Πεγιόν και τους ε, υπόλοιπους ευρωβουλευτές που τάχθηκαν υπέρ της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ξεκινήσω με τις δημοσιονομικές πτυχές των τροπολογιών του κυρίου Πεγιόν. Συμφωνώ μαζί του ως προς το θέμα της ε, ε πρό, πρόθεσης ε, νέας προσοχής, νέας εστίασης ε, των εγγυήσεων και ε, καταμέτρησης του κινδύνου των ε, διαφόρων επεμβάσεων. Σε ό,τι αφορά την αύξηση του κατοφλίου του ανώτατου ορίου θα πρέπει να δούμε τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στον ε, κοινοτικό προπολογισμό. γιατί έχουμε και τις επόμενε δημοσιονομικέ προοπτικέ και θα πρέπει να δούμε τον αντίκτυπο που θα έχει σε αυτές. Σε ό,τι αφορά τη μείωση του φέμι πρίφλο πολύ καλή πρόταση, αφορά την ευρωπαϊκή και όμως διαφορετική νομική βάση. Γι' αυτό εκεί θα μπορούσε να μας βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξεφύγουμε από το διέξοδο λόγω της διαφοράς νομικής βάσης. Ό,τι αφορά το θέμα των μικροπιστώσεων, αν αυτή η νέα εντολή προϋποθέτει μείωση των υπαρχόντων κονδυλίων και ανώτατων ορίων, γιατί το, το Συμβούλιο δεν θέλει να μειώσει τα ανώτατα όρια, ίσως υπάρξουν επιφυλάξεις για την νέα εντολή. Αν όμως προσδιορίσουμε ότι περιλαμβάνεται και η δυνατότητα κάποιων επιχειρήσεων μικροπιστώσεων θα ήταν μια πρόσδεκτη προσθήκη στην εντολή. Στα, σε ό,τι αφορά τα θεσμικά ζητήματα, για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε μια διαδικασία προβληματισμού και εξέτασης και χαίρομαι για την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά δεν θα ήμασταν υπέρα διεξοδικών διατυπώσεων όπως θέμα ε, σχετισμού ΕΤΕΠ και ΜΠΕΡΤ Γιατί μία πολύ εδελεχής διατύπωση ίσως προεξοφλήσει η ε, προδικάσεις στο μέλλον των συζητήσεων. Κάτι που απευχόμαστε. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Ντομινίκ Δεκραϊανκούρ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την Επιτροπή σας για το ενδιαφέρον που δείχνει για την πρόταση αυτή για, το για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Βεβαίω, καλωσορίζουμε το ενδιαφέρον σα αυτό, γιατί φυσικά υποστηρίζουμε πλήρω και την πρόταση τη ε, Κομισιόν. Ε, θα ήθελα όμω να ξεκινήσω λέγοντα ότι όλε οι δραστηριότητέ μα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Ε, αυτό είναι ο λόγο ύπαρξη τη τράπεζα. Και αυτό ακριβώ είναι αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε. Ότι το γεγονό ότι είμαστε εδώ σήμερα και το γεγονό ότι ο πρόεδρο Μέστατ σήμερα το πρωί έκανε την συνάντηση με του συζητητέ των πέντε επιτροπών του Κοινοβουλίου για να συζητήσει την πρόταση αυτή, δείχνει ακριβώ τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να είμαστε σε συνεχή διάλογο με το Κοινοβούλιο και θέλουμε να είμαστε και υπόλογοι στο Κοινοβούλιο όταν εφαρμόζουμε τέτοιε πολιτικέ. Για το θέμα λοιπόν αυτό, θα ήθελα να πω ότι είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία και με το Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο και με το Ελεκτικό Συνέδριο που έχει πλήρη πρόσβαση στις δικές μας επιχειρήσεις όταν μιλούμε για ε, χρηματοδοτήσεις και επίσης για τις λεπτομερείς συμφωνίες που έχουμε με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για διάφορες δράσεις που έχουν γίνει και επιτυχώς μέχρι τώρα. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που ήθελα να αφήξω. Ε, ενεργοποιούμαστε και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υποστηρίξουμε όμως τις ευρωπαϊκές πολιτικές και την ε, υπηρεσία εξωτερικών ε, υπηρεσιών. Ε, επίσης, η σύνθεση από ό,τι φαίνεται επιτυγχάνεται σιγά σιγά. Ε, δεν θα πρέπει να θεωρεί κάποιο ότι μπορεί να μετατραπεί η τράπεζα επενδύσεων σε μια αναπτυξιακή τράπεζα σήμερα. Αλλά ότι θα υπάρχει για να ε, υποστηρίξει τον χαρακτήρα των, δραστηριοτήτων της ε, ΕΤΕΠ. Αυτή είναι η ρεαλιστική προσέγγιση που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Απλώς θέλουμε να ευστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι η ΕΤΕΠ είναι ένα, ε, ένας οργανισμός με πολύ ε, λίγο προσωπικό και με αυξημένη πειθαρχία ε, στις δραστηριότητέ μας και φυσικά θα χρειαστούμε ενίσχυση σε ό,τι αφορά το προσωπικό μας για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις δραστηριότητε που κάνουμε για την απαλήψη της φτώχειας για να υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση σε επιδοτήσεις ή σε δάνεια γιατί υπάρχουν πολλές φτωχές χώρες που δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε συνθήκες αγοράς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα νόφλια, τα όρια, τα ποσά που είναι ένα θέμα σημαντικό που σας απασχολεί, φυσικά υπάρχει πρόβλημα που προκύπτει από το γεγονός ότι απαντώντας και στο δικό σας αίτημα και, στο, και, στο συμβουλίου, αίτημα του Συμβουλίου, η ε, τράπεζα έχει, ε, έχει δώσει βάρος ε, στις δραστηριότητες για να, για να απαντήσει στο αίτημα αυτό. αυτό σημαίνει όμως ότι καταναλώνονται τα ποσά πολύ, πολύ πιο γρήγορα και δημιουργείται χάσμα, δημιουργείται κενό. Πώς θα λυθεί αυτό δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Αλλά θα ήθελα να υποστηρίξω και τις ιδέες που εκφράζονται από την εισηγητή από τη... και από μέλη του Κοινοβουλίου για να μελετήσουμε κάποιους, ε, κάποιους τομείς. Ε, ίσως ας πούμε μια αναλογική αύξηση για κάποιες χώρες. Ε, ή μια άλλη λύση είναι η χρήση των ροών για τέτοιες δραστηριότητες ακόμη και αν δεν βρίσκονται μέσα σε ένα πολύ στενό προπολογισμό. Επίση, ευελιξία από μια περιφέρεια σε άλλη, σε περίπτωση, μια άλλη, κάποια, σε περίπτωση που μια ε, περιφέρεια έχει πλεόνασμα και μια άλλη έχει έλλειμμα. Ε, αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να τα, να τα δούμε. Επίσης, θα θέλω να τονίσω ότι σε ό,τι αφορά το ε, οικονομικό κέντρο, η ΕΤΕΠ έχει αναλάβει τον ηγετικό ρόλο και αυτό βεβαίω έχει αναγνωριστεί και από το Συμβούλιο ε, Κοφίν. Είμαστε οι πρώτοι ε, εναντί όλων των υπολείπων οικονομικών ε, ιδρυμάτων και αυτό βεβαίω ε, δημιουργεί και κάποιε δυσκολίε. Γιατί εμεί έχουμε και πολύ αυστηρέ ε, πολιτικέ. και αυτό βεβαίω δεν διευκολύνει τη δουλειά μα. Και κλείνοντα να πω ότι τα θεσμικά θέματα είναι επίση πολύ δύσκολα και περίπλοκα και μάλλον δεν θα ήταν φρόνιμο να, το, να τα λύσουμε τώρα, ε, στα πλαίσια και της ενδιάμεσης δηλαδή αξιολόγησης, αλλά ίσως ε, στα πλαίσια της επόμενης εντολής. Εν τω μεταξύ βεβαίως είμαστε απολύτως αφοσιωμένοι στο να δημιουργήσουμε πλατφόρμες συνεργασίας, όπως προτείνεται από, την, ε, από τον εισηγητή σας, με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Αλαφράγκα ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που παρεμβαίνω τόσο αργά στη συζήτηση. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Πεγιόν για την ε, έκθεσή του, για το σχέδιο έκθεσής του και όπως είπαμε ε, υπάρχει ε, μία ειδική πτυχή εξωτερικής δράσης, γιατί ακριβώς το 10% των το χρηματοδοτήσεων απευθύνονται σε συνεργάτες, σε συνεργασίες Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες και γι' αυτό και ε, έτσι διαφαίνεται ο ρόλος της ΕΤΕΠ ε, όσον αφορά τη στήριξη της ανάπτυξης. Θα πρέπει να προσέξουμε ωστόσο πάρα πολύ χρησιμοποιώντας τους πόρους που μας δίνει η εξωτερική μας πολιτική και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε να συντονιστούν όλα αυτά με την Επιτροπή και με τις υπηρεσίες της ΥΠΑ της εκπροσώπους. Έχουμε διάφορα μέσα, το προενταξιακό μέσο, τα η πολιτική ε, γυτνίασης ε, της ε, Βραζι... Βραζιλία, Κίνα, Μεξικό κτλ. Η συνεργασία με διάφορους οργανισμούς κρατών της Λατινικής Αμερικής και ούτω, ούτω, καθεξής. Ωστόσο, θα πρέπει να δούμε ποιε, και ποιε θα είναι οι νέες δημοσιονομικές προοπτικές της Ένωσης και οι γεωγραφικές ισορροπίες που θα συσπιστούν μέσα στο πελαίσιο αυτό θα πρέπει να τα διαπραγματευτούμε, να τα διατυπώσουμε επί τη βάση των συμβιβαστικών λύσεων που έχουμε ήδη ε, συμφωνήσει. Και νομίζω πως αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη γιατί είναι πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα. <coughs> Πριν να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Πεγιών για να ολοκληρώσει. Θα ήθελα προσωπικά να τον συγχαρώ για την εξαίρετη του εργασία που βρίσκω πολύ ισορροπημένη. Παρακαλώ κύριε Πεγιών. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ όλους Καταρχήν να ε, Ευχαριστήσω τον συνάδελφο Σαλαφράγκα για την έκκληση σε σύνεση που μας έκανε και άλλοι συνάδελφοι το είπαν. Ε, καταλαβαίνουμε ποια είναι η εξαιρετική περιπλοκότητα αυτής της ε, υπόθεσης και η κυρία Γιαννάκου είπε κάτι πολύ σωστό και το οποίο μπορούμε να τονίσουμε περισσότερο στην έκθεση αν το επιθυμείτε, αλλά που στην ουσία αποτέλεσε το νήμα της ε, Αριάδνης για αυτήν εδώ την έκθεση να δούμε δηλαδή ποιος είναι ο πραγματικά ο στόχος όλων αυτών, διότι πρέπει να συνδυάσουμε από τη μια πλευρά την αναπτυξιακή βοήθεια, την πολιτική ε, ανάπτυξη και τα ακούσαμε για τις φτώχειες χώρες, αλλά και να στηρίξουμε τα συμφέροντα, τα οικονομικά της Ένωσης σε μέρη όπου έχουμε ανταγωνιστές και όπου δεν πρέπει να είμαστε αγαθοί και να μην έχουμε μέσα παρέμβαση στη διάθεσή μας. Αυτές οι δύο λογικές ε, βεβαίως μπορούν να ενταχθούν σε μια απόλυτη συνοχή, αλλά και κάποιες φορές μπορεί και να έρθουν σε σύγκρουση. Άρα λοιπόν θα πρέπει ταυτόχρονα να ανταποκριθούμε στους στόχους, της πολιτικής της Ένωσης ε, όσον αφορά την ανάπτυξη και ταυτόχρονα την οικονομική και δημοσιονομική ισχύ της Ένωσης σε έναν κόσμο όπως έχει σήμερα, τελείως ανοιχτό, όπου και ακόμα και στις χώρες της υποανάπτυξη υπάρχουν από άλλε μεγάλες χώρες που ε, παίζουν ανταγωνιστικό σε εμά ρόλο. Και έπειτα κύριε Γεννάκου για την ερώτηση, τον προβληματισμό του κατά πόσο είναι βανάγνωστες οι πολιτικές ανάπτυξη μας. Το συζητήσαμε πρόσφατα όσον αφορά την Μέση και η Εγγύης Ανατολή. Η Ένωση έχει πολύ περισσότερα χρήματα από όλους τους άλλους, αλλά αυτό δεν είναι πάντα ορατό. Δεν είναι πάντα ορατό και ούτε και το πολιτικό μας κύρος αντισταθμίζεται και μάλλον ανταμείβεται από αυτή την άποψη. Το έχουμε υπόψη μας λοιπόν κυρία Γιαννάκου, να ανησυχείτε. Τώρα βεβαίως και είναι ένα από τα στοιχεία της έκθεσης κυρία Όταλα, δηλαδή προσπάθεια διαφάνειας. Ναι, πρέπει να είναι μόνιμη η προσπάθεια αυτή και διαρκής. Αυτό ήδη εντάσσεται στη βούληση καλύτερο συντονισμό, μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ της Κομισιόν και των χωρών, στις προσπάθειες που κάνει η ΕΤΕΠ για να ενημερώνει για τις δραστηριότητές της και εμείς στο Ευρωκοινοβούλιο ζητούμε ακόμη περισσότερο για τις μικροπιστώσεις. Δεν είναι μόνο πόσα που προσπαθούμε να προσθέσουμε, ούτε για τι αυξήσει που σα είπα για τι πέντε νέε χώρε. Είναι διαδικασίε τι οποίε προσπαθούμε να καταστήσουμε πιο αποτελεσματικέ. ενισχύοντας τη συνεργασία, εν, βρίσκοντας έναν χώρο για την εξωτερική υπηρεσία και σε πλήρη και διαρκή συνεργασία και με το Κοινοβούλιο. Δεν θέλουμε να είμαστε ένα απλά εκτελεστικό όργανο. Κάνουμε ολόκληρη δουλειά εδώ και τα λέω αυτά και για το συνάδελφο Χουντή. Ε, δεν θα δίνουμε απλέ εγκρίσει. Νομίζω πω ο διαχωρισμό των εξουσιών είναι μέγα κεκτημένο τη δυτική δημοκρατία και το διατηρούμε φυσικά. Ε, αντίθετα και νομίζω ότι εδώ σωστά έχουμε βρει μια συνένεση και υπάρχουν ήδη αιτήματα για τα δύο δις επιπλέον όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές. Και για να ολοκληρώσω και όλες οι ανησυχίες που εκφράσατε κυρία Όταλα και κυρία Γιαννάκου θεωρώ πως είναι θετικές. Να απαντήσω στον κύριο Σαλαβράκο για να ολοκληρώσω. Ας προσέξουμε πολύ οι δημοσιονομικές δυσκολίες που μπορεί να ε, συναντούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες μέλη να μην μας οδηγήσουν στο να περιορίσουμε τις εξωτερικές μας πολιτικές. Γιατί το μέσο οικονομικής ανάπτυξης φυσικά βασίζεται μέσα στην Ένωση αλλά και εκτός αυτής και αν οι αποφάσεις μας ε, ε συνίστανται στο να μην παίξουμε πλέον ε, ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη τότε θα απομονωθούμε και θα χάσουμε ένα μεγάλο οικονομικό πλεονέκτημα. Ναι, εντάξει, υπάρχουν δυσκολίε, αλλά να μην εγκαταλείψουμε ένα σωρό όπου υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχουν ανάγκες, όπου μπορούν να βρίσκονται οι εταιρείε μας και όπου η ανάπτυξη και η καταπολέμηση της στόχης και εσείς κυρία Ότελα το προσθέσατε η υγεία και η ε, παιδεία, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά τα δικά μας μέσα για την ανάπτυξη των αξιών μας, αλλά και για την οικονομική ανάπτυξη. Ε, αν δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητέ, να περάσουμε στο τελευταίο σημείο τη ε, πρωινή συνεδρίαση, η εξέταση τη έκθεση ε, του συναδέλφου Μπέλντερ για την συνεργασία, την προσέγγιση μάλλον της Ένωσης προς το Ιράν. Πολύ ανησυχητική κατάσταση όσον αφορά την εσωτερική πολιτική και την πυρηνική ενέργεια που δεν έχουν υπάρξει πρόοδοι παρά τις διάφορες προσπάθειες που έχει καταβάλει η διεθνής κοινότητα, η Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία από την μια πλευρά, ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία από την άλλη το ψήφισμα 1929 που υιοθετήθηκε από τον Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 9 Ιουνίου 2010 επέβαλε μια τέταρτη, ένα τέταρτο γύρο κυρώσεων στο Ιράν που συνοδεύτηκαν από κυρώσεις που αυτόνομα επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΙΠΑ, η Ιαπωνία, ο Καναδάς και η Αυστραλία. Η έκθεση του κ. Μπέλντερ που θα συζητήσουμε σήμερα εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο αυτό και ε, μας έρχεται σε μια πολύ ευαίσθητη φάση των σχέσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ιράν. Να θυμίσω εν τέλει ότι η επίσκεψη στο Ιράν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ε, ναι, από την αντιπροσωπεία για το Ιράν, συνεργασία μάλλον με το Ιράν, στι οποίε ηγήθηκε η κυρία Λόχ Ντίλερ, που είναι παρούσα, ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή από πλευρά των Ιρανικών αρχών. Παραμένουν λοιπόν αμφιβολίες για το τι ακριβώς συμβαίνει και για το αν θα μπορέσουμε, τελικά, αν τελικά θα μπορέσει να γίνει αυτή η επίσκεψη. Θα δώσω λοιπόν το λόγο αυτή τη στιγμή στον κύριο Μπέλτερ για την παρέμβασή του. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι. Μετά από ενδελεχή μελέτη, θα ήθελα πολύ σύντομα να σας αναφέρω κάποια πράγματα για τη γνωμοδότησή μου. Έπρεπε να διαγράψω σχεδόν τη μισή μου γνωμοδότηση για να είναι έτσι πιο συνεπτυγμένη, για να δείξω ποιε είναι οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιράν. Ε, συμμερίζομαι ε, και, και για λόγο διαφάνειας ότι... Ε, έχουμε τα κεφάλαια, τα κεφάλαια για την ιστορική κατάσταση, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το πυρηνικό πρόγραμμα και το αντίστοιχο πρόβλημα που προκύπτει και οι εξωτερικές σχέσεις του Ιράν. Για την εσωτερική κατάσταση τώρα στη χώρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ιρανική κυβέρνηση πραγματικά βρίσκεται ενώπιον σημαντικών προκλήσεων. Υπάρχει μεγάλη ναι, διαμάχη μεταξύ επαναστατικών φραξιών στη χώρα για κοινωνικά και οικονομικά θέματα. Η κατάσταση επιδεινώνεται δυστυχώς ε, συνέχεια ε, και αυτό βεβαίως έχει ε, συνέπειες και στον πληθυσμό ο οποίος γίνεται όλο και λιγότερο υπομανετικός. Βεβαίως θα πρέπει και η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα δυναμικά, τα προβλήματα που ε, προκύπτουν μετά τις ε, νικηφόρες ε, προεδρικές εκλογές. Ο πρόεδρος Αχμαντινετζάντ μίλησε στεναρά για την Ισλαμική Επανάσταση. Εγώ θα ήθελα στην, σε σχέση με αυτό να σας θυμίσω ότι υπάρχει και ένα ε, κινηματογραφικό έργο το οποίο παρουσιάζει πάρα πολύ καλά αυτή την ε, κατάσταση. Νομίζω το λένε το πράσινο κύμα. Ε, τώρα, για, την, για τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας και την κοινωνική γενικώ κατάσταση η χάρτα για την Ισλαμική Επανάσταση προκύπτει, μάλλον μετατρέπεται σε ένα κράτο εν κράτη. Η σχετική, το σχετικό κίνημα μετά τα αποτελέσματα της, ε, των εκλογών ξεκίνησε μια διαδήλωση λέγοντας ε, πού είναι η δική μου η ψήφος. τώρα ρωτούν πού βρίσκονται τα, πού πάνε τα λεφτά από το πετρέλαιο και αυτό είναι σημαντικό. Ε, τώρα πάμε στα ανθρώπινα δικαιώματα. Σαφή παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως πάντα στην ε, χώρα αυτή. Ε, παρατηρούνται πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα. Και βεβαίως ε, εγώ θα ζητούσα να απαιτήσουμε το εξή. Η Κομισιόν και το Συμβούλιο να δώσουν έναν κατάλογο στον, ε, στο Ιράν με συγκεκριμένα παραβιάσεις που έχουν παρατηρηθεί και να απαιτήσουν να γίνει έρευνα. Να υπάρξουν ευθύνε, να υπάρξουν συλλήψεις, να γίνει δίωξη. Δεύτερον, πρέπει να πιεστεί η Ιρανική κυβέρνηση, γενικώ οι Ιρανικές αρχές, επιτέλους να αφήσουν να μπουν στη χώρα οι εκπρόσωποι απεσταλμένοι το ΟΗΕ. Επίσης, κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι όσους είναι ακτιβιστές ε, και δραστηριοποιούνται στην, στο Ιράν να τους ενισχύσουμε γιατί πραγματικά και αυτοί υπόκεινται ε, πάρα πολλά. Ε, επίσης θέμα ελευθερίας των ε, θρησκευτικών πεπιθήσεων. σε επίσημες επισκέψεις στο Ιράν βλέπουμε πάντα λίστες με άτομα που έπεσαν θύματα καταπάτησης δικαιωμάτων, πολιτικοί κρατούμενοι που πρέπει να ελευθερωθούν. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα και είναι πολύ συγκεκριμένα. Πρέπει λοιπόν να, στα συγκεκριμένα, επί των συγκεκριμένων να επικεντρωθούμε και να δράσουμε. Πέρα από αυτό, Πρέπει και η ιρανική μπλογκόσφαιρα να ε, ενισχυθεί όπως λέμε σήμερα γιατί νομίζω ότι και αυτή έχει κάνει πάρα πολύ, ε, καλό, πάρα πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια. Κάτι άλλο. Οι επαφές μεταξύ βουλευτών και του δικού μας, μεταξύ του δικού μας κοινοβουλίου και του Ιρανικού θα πρέπει να βελτιωθούν φυσικά οι σχέσεις μας. Βεβαίως θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην κατάσταση, στις συνθήκες κατά από τις οποίες ζουν οι άνθρωποι στο Ιράν. Πρέπει να πούμε ότι το Ιράν εμποδίζει την ε, διεθνή ε, υπηρεσία ε, πυρηνικής ενέργειας να κάνει τη δουλειά της. Το Συμβούλιο θέλει να εξεύρει μια ε, καλή λύση μεν, αλλά θέλει να ζητήσει και από την... Θέλει να... Πρέπει να δούμε και ποια είναι η κοινή θέση του Συμβουλίου ήδη από τον Ιούλιο του 2006 και κατά πόσο αυτή εφαρμόζεται και γίνεται σεβαστή. Και επίσης ε, και το Συμβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει ε, να συμφωνήσουν επί μιας πολιτικής και με τις ΗΠΑ για τα θέματα ανθρώπινων ε, δικαιωμάτων και αξιοπρεπούς μεταχείρισης. Το Ιράν απειλεί την ε, Ανατολή, την σταθερότητα στην περιοχή θέλει να επηρεάσει τα πράγματα ώστε να απορριθμιστεί η κατάσταση σε όλη αυτή την περιοχή. Και είναι αξιοπρόσεκτο πώς εξελίσσονται οι σχέσεις του Ιράν και με την Τουρκία και πώς έχουν αλλάξει. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης θα πρέπει να ε, μιλήσουν με συγκεκριμένη φωνή και προς την Τουρκία και να ζητήσουν να ενισχυθεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου Τώρα, σε ό,τι αφορά το, του, ε, το πάγιο αίτημα του, ε, του Ιράν να εξαφανιστεί από τον χάρτη το Ισραήλ. θα πρέπει να δούμε το θέμα αυτό. Ε, θα πρέπει να έρθουμε με μια συγκεκριμένη πρόταση και ως προς αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και βεβαίως προσβλέπω στις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ. Τώρα. Ε, πρόεδρος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Ιράν, η κυρία Λόχ Παρακαλώ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπέλτερ για την έκθεση. Καταρχήν να πω ότι Χτες λάβαμε την γραπτή εκδοχή του, της εκθεσής του, οπότε ε, έτσι παρατηρήσεις εν είναι αυτές που θα ακούσετε σήμερα και επίσης η προθεσμία για την ε, υποβολή τροπολογιών είναι η 12η Οκτωβρίου. Είναι πάρα πολύ στενά τα περιθώρια που μας δίνονται είναι η πρώτη ε, ας πούμε, απόπειρα που κάνουμε για το θέμα του Ιράν και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να έχει αρκετό χρόνο για να συζητηθεί. Ε, είναι λίγο στενά τα περιθώρια που μας δίνεται, εν πάση περιπτώσει. Ε, θεωρώ ότι είναι πολύ σωστό ο τρόπος με τον οποίο έχει διαρθρώσει την γνωμοδότησή του ο κ. Μπέλντερ. Μιλούμε για τον ρόλο του Ιράν στην ευρύτερη ναι. περιοχή. Και δεν μιλούμε μόνο για τις αρνητικές επιπτώσεις και για τις συνέπειες, για τις απειλές του Ιράν, αλλά θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να υπάρξει συνεργασία. Θεωρεί ότι η συνεργασία είναι απαραίτητη με το Ιράν ε, όταν μιλούμε για την κατάσταση ας πούμε στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Επίσης σημαντικό είναι να υπάρξει μια συνολική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι του Ιράν. Να μην μιλούμε δηλαδή μόνο και με μονομένε πτυχέ και να τις καταγράφουμε, αλλά να υπάρχει σε μια σύγκληση όλων αυτών. Φυσικά είναι αυτονόητο ότι η διεθνής πολιτική βρήθη των ε, παραδειγμάτων από σχέσεις πολιτικές μεταξύ ΙΠΑ και Ιράν, αλλά νομίζω ότι η παρούσα κυβέρνηση των ε, ΙΠΑ έχει επιλέξει μία προσέγγιση που προωθεί τις πολιτικές λύσεις. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουμε μία δική μας μεμονωμένη πολιτική για το Ιράν. Βεβαίως και σε συμφωνία με τις ΗΠΑ κατά πάσα πιθανότητα. Επίσης, χαιρετίζω το γεγονό ότι αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις που κατέρευσαν τελικά μεταξύ Βραζιλίας και Τουρκίας ε, να μην ε, αναφέρονται στην γνωμοδότηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε όμως μια θετική χρειά όλο αυτό. Ότι δηλαδή ο διπλωματικός ρόλος της Τουρκίας για την Ευρώπη θα μπορούσε να είναι σημαντικός θα μπορούσαμε ο ένας να ενισχύσει τον άλλον ώστε να υπάρξει τελικά αυτή η πολιτική λύση που όλοι επιθυμούμε. Τώρα, για τα μεμονωμένα επιμέρους ερωτήματα. μπορώ να σας δώσω τις απαντήσεις μου για τον κάθε τομέα, δηλαδή γραπτός καλύτερα, αλλά πέρσι από τότε που άρχισε, που ξεκίνησε η ε, θητεία μας, έχουμε τρεις, ε, τρία ψηφίσματα για το ε, Ιράν. τα, για, τα οποία όμως περιλαμβάνουν ε, διαφορετικά, ε, διαφορετικές απαιτήσεις. Ας πούμε υπάρχουν, ε, υπάρχει η μακροπρόθεσμη ε, προσέγγιση για, την, για να υπάρχει ελευθερία από πυρηνικά όπλα στην περιοχή. Επίσης να συμπληρώσω κάτι, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γνωμοδοτούν είτε επίσημα είτε ανεπίσημα. Έχουμε και την ε, αντιπροσωπεία για το Ιράν για να βλέπουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις που υπάρχουν ε, μετά τις ε, κυρώσεις που επιβάλλονται στο Ιράν. Θα μπορούσαμε λοιπόν ε, ίσως να συμπεριλάβουμε στη γνωμοδότηση μια παράγραφο που θα λέει ότι θα υπάρχει σε τακτικά χρονικά διαστήματα μια έκθεση από την Κομισιόν βεβαίως σε ε, συμφωνία με την ε, αντίστοιχη Επιτροπή Κυρώσεων του ΟΗΕ. Να δούμε δηλαδή ποιε είναι οι κυρώσει που επιβλήθηκαν, αν όντω εφαρμόστηκαν, αν όντω είχαν αποτέλεσμα. Τώρα για τον φάκελο για τα πυρηνικά, να δούμε κατά πόσο οι κυρώσει αυτέ έχουν επίση συνέπεια συγγνώμη, στην στην κοινή γνώμη. Επίσης, παράγραφος 14. Μιλούμε για την ε, αντιπροσωπεία του Ιράν και για, την, ε, για, τις, για, τους, ε, για τις προαιρέσεις που υπάρχουν για τις επισκέψεις προς το Ιράν. Ε, νομίζω ότι αυτή είναι άδικη μεταχείριση έναντι άλλων αντιπροσωπιών, ε, γιατί δεν μπορούμε να λέμε ότι αν υπάρχουν συγκεκριμένε αλλαγέ ε, έναντι των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μόνο τότε θα ταξιδέψουμε στη χώρα. Νομίζω ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Δεν μπορούμε να δείχνουμε τέτοια δείγματα στι γειτονικέ χώρε, στην Κίνα, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ. Νομίζω ότι αυτό, αυτή είναι η λαθασμένη προσέγγιση. Και τέλος, να πω το είπε βεβαίω και ο κ. Μπέλγκαρ στα αρχικά του σχόλια, ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ε, θέση στην οποία βρίσκεται η πολιτική, ε, η αντιπολίτευση στη χώρα είναι πραγματικά δεινή. Δεν έχει υπάρξει καμία βελτίωση, πραγματικά καμία. Και αυτή η εσωτερική κατάσταση έτσι όπως εξελίσσεται οφείλεται ακριβώς στην, ε, στις δράσεις της κυβέρνησης. Ε, υπάρχουν πολλοί στην, ε, στον ιρανικό πληθυσμό που υποφέρουν από αυτή την κυβέρνηση. Θεωρώ λοιπόν ότι σκόπιμο θα ήταν στην γνωμοδότησή μας να έχουμε ένα σημείο το οποίο θα μιλά για τη σημασία της χώρας, για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων κάτω από την κυριαρχία του, της σημερινής κυβέρνησης έτσι ώστε να έχουμε μια γρομοδότηση η οποία θα έχει μια μεγαλύτερη ε, διάρκεια και θα δείχνει ποια είναι η σαφή θέση του ε, Κοινοβουλίου. Πρέπει να μιλήσουμε για, την, ε, για, τον, για το πυρηνικό φάκελο, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τις παραβάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, για τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η πολιτική που ακολουθεί το Ιράν στην περιφέρεια, αλλά θα πρέπει πάντα να διαχωρίζουμε γιατί, τα πράγματα γιατί η κυβέρνηση ακολουθεί μία άγουσα αλλά οι πολίτες πολύ συχνά έχουν τελείω διαφορετική άποψη. Ευχαριστώ. Μάλιστα, πριν δώσω το λόγο στη συνάδελφο Μονής που είναι σκιώδης εισηγήτρια των σοσιαλιστών να σας πω ότι η διορία για την υποβολή των τροπολογιών είναι 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Όπως σας είχαμε πει και χτες, μα μήπως, νομίζω πως δεν το γνώριζαν όλοι. Νέα διορία λοιπόν, 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. κυρία Μουνής. Σας ευχαριστώ. Έχουμε εγκρίνει πληθώρα ψηφισμάτων για διάφορες πτυχές ε, της ιρανικής πολιτικής. Ήδη εγκαινιάσαμε τη θητεία μας με τρία νέα ψηφίσματα. Έχουμε διοργανώσει ένα σωρό συνδιασκέψεις, σεμινάρια. Έχουμε καταρτήσει μελέτες για το Ιράν και το σημαντικό του ρόλο ως περιφερειακού και παγκόσμιου εταίρου. Γιατί έχει και γεωστρατηγική θέση. Έχουμε επιτέλου την ευκαιρία να συντάξουμε και μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα είναι σημείο αναφορά τη ευρωπαϊκή πολιτική προ το Ιράν. Θα χρειαζόμαστε ένα συνολικό πλαίσιο και μια συνολική ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στο Ιράν. Δεν θέλουμε μια έκθεση φυσικά που είναι τελείως αντιφατική με προηγούμενες θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό θα πρέπει να έχουμε συνείδηση κατά την κατάρτιση αυτής της έκθεσης. Ο κύριος Μπέλντερ εκπώνησε ένα σχέδιο έκθεσης με αρκετά ενδιαφέρουσα δομή, αλλά με σημαντικές ελλείψεις ως προς το περιεχόμενο. Τα πιο σημαντικά θέματα, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, επικεντρώνεται κυρίως στη δίωξη των ε, θρησκευτικών μειονοτήτων. Αλλά δεν γίνεται λόγος ούτε για τις γυναίκες, για την καταπίεση που υφίσταται οι γυναίκες, δεν αναφέρονται οι ομοφιλόφιλοι, δεν, αναφέρονται, ε, δεν αναφέρεται η θανατική ποινή, η δίωξη ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατάφαρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά τα θέματα δεν, δεν αναφέρονται. Μία έκθεση για το Ιράν που έχει κεφάλαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορεί να είναι πλήρη εφόσον ε, δεν αναφέρει τα πιο σημαντικά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απασχόλησαν κατά καιρό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί επικεντρώνονται μόνο στι θρησκευτικέ μειονότητε. Επίση, για τα πυρηνικά θέματα δεν αναφέρονται οι τελευταίε εξελίξει, δηλαδή η προσφορά τη Τουρκία και τη Βραζιλία και οι επιπτώσει που μπορεί να προκύψουν από αυτέ τι νέε εξελίξει. Δεν γίνεται λόγο για τα θέματα αυτά. Σε ό,τι αφορά τι εξωτερικέ σχέσει και πάλι επικεντρώνεται τη έκθεση σε ένα μόνο θέμα, το θέμα του Ισραήλ. Ούτε συμφωνώ με την θέση που εστερνίζεται για την Τουρκία ο κύριος Μπέλτερ. Η Τουρκία όντως είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη θέση της χώρας αυτής αλλά και τις σχέσεις της με το Ιράν. Γιατί το Ιράν είναι περιφερειακό παράγοντα, αλλά οι σχέσει με την Τουρκία δεν αποσταθεροποιούν αυτή την κατάσταση, αλλά μάλλον την σταθεροποιούν. Ούτε αναφέρεται ο ρόλο του Ιράν σε σχέση με το Αφγανιστάν, την Κεντρική Ασία και ο θεμελιώδη ρόλο του Ιράν στο Αφγανιστάν μετά την διαμάχη με τους Ταλιμπάν, γιατί εκεί διαδραμάτισε θεμελιώδη ρόλο το Ιράν. Κάτι άλλο που λείπει από την έκθεση Belder που έχει όπως είπα σωστή δομή λείπει ένα κεφάλαιο με προτάσεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ιράν. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Μεταναστευτική πολιτική. Στην Τουρκία 6.000 ε, Ιρανοί πρόσφυγες περιμένουν να, ε, ε, να φύγουν προς την Ευρώπη. Και υπάρχουν κάποιες προτάσεις διμερείς με τη Γερμανία και την ε, Ολλανδία. Γιατί να μην προτείνουμε μια πανευρωπαϊκή πολιτική μεταναστευτική ή επίλυση του προβλήματος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για αυτούς τους πρόσφυγες. Η κυρία Λόχμπιλερ ανέφερε το σημείο 14 που εξαρτά την ε, δυνατότητα πραγματοποίησης ε, αποστολών από τη βελτίωση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να προωθήσουμε οποιαδήποτε δυνατότητα ελέγχου, ε, ε, διαλόγου με τις Ιρανικές Αρχές και δεν μπορούμε να εξαρτούμε το διάλογο από εσωτερικές αλλαγές που μέχρι στιγμής το άλλως δεν ε, υλοποιήθηκαν. Σε ό,τι αφορά την εσωτερική κατάσταση, παρά είναι σχηματική η προσέγγιση του κυρίου Μπέλτερ, αναφέρονται μόνο οι θεματοφύλακες της Επανάστασης. Το Ιράν είναι μια χώρα με πολύ περίπλοκη, σύνθετη εσωτερική κατάσταση. Δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε στην εσωτερική μόνο η οργανωτική διάρθρωση του Ιράν. Βέβαια υπάρχουν κάποια σημεία που είναι αρκετά εύστοχα και αποδεκτά, αλλά θα πρέπει να ενισχυθούν. Το σημείο 8 για την μπλογκόσφαιρα και την προστασία των blogger. Ωραία, αλλά ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητήσαμε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με τεχνολογίες επικοινωνίες να αποφεύγουν εξαγωγή τεχνολογίες διπλής χρήσης που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από το Ιράν για την καταπίεση ή τον περιορισμό της χρήσης του διαδικτύου. Στην παράγραφο 12 αναφέρεται ε, εκπρόσωπος των ειδικών ε, εντεταλμένων το ΟΗΕ για τα θέματα του Ιράν. Εδώ ζητήσαμε ένα μόνο ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών να έχουμε με ειδική εντολή για τα θέματα του Ιράν. Και μάλιστα το είχαμε ήδη το 2020. Γιατί να μην επανέλθουμε σε αυτή την κατάσταση. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε εγκρίνει διάφορα ψηφίσματα. Θα πρέπει λοιπόν να συμπληρώσουμε πολλές παραγράφους και να επανισορροπήσουμε την έκθεση. Και όταν μιλούμε για ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε μόνο στην δίωξη των θρησκευτικών κοινοτήτων. Θα πρέπει να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής γιατί και άλλα ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων υπάρχουν στο Ιράν και όχι μόνο των θρησκευτικών μειονοτήτων. Το τελευταίο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε κυρώσεις κατά των ε, αυτούργων παραβίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Πρόσφατα το έκαναν και οι Ηνωμένες και το ζητήσαμε και εμείς από το Συμβούλιο. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να περιληφθούν στην έκθεση. Πολλές βελτιώσεις λοιπόν θα πρέπει να περιληφθούν στην έκθεση και χαίρομαι για την παράταση της προθεσμίας για την κατάθεση των απολογιών. Αυτά και ευχαριστώ τον κύριο Μπέλτερ για την έκθεσή του. Το λόγο τώρα έχει ο άλλος και ηγητής, ο κύριος Γκάλερ. Ελκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους, τον κύριο Μπέλτερ για την έκθεσή του και βεβαίως οι συνάδελφοι που μίλησαν ήδη, είπαν πολλά από αυτά που ήθελα να πω εγώ, θέματα για την δομή, φυσικά είναι πολύ σωστά. Ε, οι συνάδελφοι επίσης ανέφεραν και κάποια σημεία ε, τα οποία με απασχολούσαν για μένα, οπότε δεν θα χρειαστεί τώρα να τα επαναλάβω. Η σχέση τώρα μεταξύ ε, εδαφίων και παραγράφων. Ε, υπάρχουν πολλές παύλες, πολλά έτσι μικρά εδάφια στην έκθεση τα οποία νομίζω θα μπορούσαν να συγχωνευτούν σε μια μεγάλη παράγραφο ή δύο, εν πάση περιπτώσει να υπάρχουν έτσι συγκεκριμένα θέματα. τώρα για τη δήλωση της κυρίας Άστον, ίσως θα μπορούσαμε πιο λεπτομερέστερα να την έχουμε συμπεριλάβει. τώρα νομίζω ότι για τον ε, τομέα της εσωτερικής πολιτικής, που επίσης αναφέρθηκε εν μέρη, για να καταλάβει κανείς το Ιράν, θα πρέπει να ορίσει ποιοι είναι οι βασικοί φορείς. Είναι ούτω ή άλλω από, απ' έξω να αξιολογήσουμε εμεί πώ γίνεται η αλλω δυσκολο απο απ εξω να αξιολογησουμε πληροφοριών και ποιε είναι οι δομές που ανταλλάσσουν πληροφορίες και συνεργάζονται και λαμβάνουν αποφάσεις. Σίγουρα όμως πρέπει τους βασικούς παίκτε να του αναφέρουμε. Το, το Συμβούλιο Expedency, το, την, ε, το Assembly of Experts, ε, τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων και άλλους, εν πάση περιπτώσει, σημαντικούς φορείς οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις. Αν δεν αναφέρονται εδώ, νομίζω ότι δεν θα είναι σωστή η αξιολόγηση που κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρίσταται με συγκεκριμένες πολιτικές, ναρκωτικά ας πούμε, έλεγχος των ναρκωτικών, στον αναπτυξιακό τομέα επίσης ε, ανθρωπιστική βοήθεια για κρατουμένους, συνεργασία που υπάρχει στον τομέα αυτό. Αυτά θα πρέπει να αναφέρονται. Εμείς ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να βελτιώσουμε την ε, πληροφόρηση που λαμβάνουμε από, την, ε, από το Ιράν. Επίσης είπαμε ότι θα, συμφωνήσαμε ότι θα, τα, τα Euronews θα ε, εκπέμπονται και, στα, και στα φαρσί. Ε, θα ξεκινήσει και αυτό να λειτουργεί. Ε, τώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά που αναφέρονται στην έκθεση είναι σωστά, αλλά θεωρώ ότι την παραβίαση των ανθρωπινών δικαιωμάτων θα πρέπει να την αναφέρουμε και για άλλους πληθυσμούς. Την αναφορά, έτσι, την αναφορά της παράβασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να την αναφέρουμε και σε σχέση με μειονότητες, θα πρέπει να αναφέρουμε την ποινή του θανάτου, την διακριτική μεταχείριση των γυναικών. αυτά θα πρέπει να αναφέρονται ρητά. Να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι και σε ό,τι αφορά την ε, απόφαση που υπάρχει για την 20ετή φυλάκιση ε, για την περίπτωση αυτή που προέκυψε πρόσφατα στο Ιράν. Ε, νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να το αφήσουμε, να μην το ξεχάσουμε, να συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση. Για τις εξωτερικές σχέσεις τώρα. Είναι σημαντικό να είναι σαφές ότι δεν μιλούμε μόνο για συνεργασία μεταξύ ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο αυτή σημαντική. Νομίζω ότι είναι επίσης σημαντικό να μιλούμε και για το παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή να μιλούμε για το επίπεδο του ΟΗΕ. Και εκεί να μπορέσουμε να καταστήσουμε σαφές στο Ιράν ότι ολόκληρη η παγκόσμια κοινότητα είναι ε, αντίθετη με το πυρηνικό του πρόγραμμα το Συμβούλιο Ασφαλείας φυσικά είναι σημαντικό. Βεβαίως υπάρχει και το δίλημα του ότι δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πολύ σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις με την Κίνα. Αλλά το να, το να μπορούμε να καθίσουμε απέναντι στο Ιράν, στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να πούμε ότι όλος ο κόσμος είναι αντίθετος με το πυρηνικό σου πρόγραμμα, αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό και θα πρέπει ρητά να αναφέρεται στην ομοδότηση και θα πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπαθίες μας έτσι ώστε να ε, υπάρξει μια κοινή θέση, μια κοινή αντιμετώπιση ε, ε, για το Ιράν. Ο συνάδελφος, είπε ένα συνάδελφος ότι ο συνάδελφος Μπέλτερ κρίνει, την, κατακρίνει μάλλον την θέση της Τουρκίας. Εντάξει, καμιά φορά είναι λίγο περίεργα αυτά που ακούγονται από την Τουρκία για το Ιράν. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ σημαντικό αυτό. Για τον πυρηνικό φάκελο θα ήθελα να το διευρύνουμε λίγο το σχετικό κεφάλαιο. και να συμπεριλάβουμε και τις εξωτερικές σχέσεις. Να συμπληρώσουμε δηλαδή όπως το πρότειναν και άλλοι συνάδελφοι. Ε, αυτά. Πρόεδρε, από μένα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η σκιώδη συγκεντρία της Γκουε, η κυρία Λέζινγκ. Ευχαριστώ. Äh, aufgrund des Zeitfensters äh, Θα ήθελα να ε, σχολιάσω λίγο αυτά που ακούστηκαν, ε, να, κάνω, να δώσω πια, τις βασικές θέσεις της ε, Γκούρας προς το συγκεκριμένο θέμα του Ιράν. Να πω καταρχήν ότι την ε, δύσκολη πολιτική κατάσταση στο Ιράν, την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση του Ιράν και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων την καταδικάζουμε ε, παρόλα αυτά, το πώ την διαχειρίζεται η έκθεση αυτή, την όλη αυτή κατάσταση, νομίζω ότι πρέπει να το επικρίνουμε ε, γιατί μιλούμε για την αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής έναντι του Ιράν, ώστε να ε, απομονώσουμε το Ιράν. Ε, να, τελειώσουν, να τελειώσει η πολιτική των κυρώσεων, ειδικά σε ό,τι αφορά τα θέματα του πυρηνικού προγράμματος, αλλά και ε, σε ό,τι αφορά την ελεύθερη ζώνη στη Μέση και Αγγής Ανατολή, ε, ελεύθερη ζώνη από πυρηνικά όπλα. Ε, επιμένουμε στην συμπερίληψη και στην επανεκκίνηση του πολιτικού διαλόγου ώστε να βρούμε μια διπλωματική και ειρηνική λύση για το Ιράν και θα επαναλάβω ότι η όξυνση των κυρώσεων σίγουρα δεν θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση θα δημιουργήσει το αντίθετο αποτέλεσμα. Είναι προφανές και αυτό το είδαμε και στο παρελθόν και έχει αποδειχτεί ότι μέσω των κυρώσεων οι φονταμεταλλιστικές θέσεις ενισχύονται και αυτό ενισχύει τη θέση του Αχμαντινετζάτ και τα προγράμματα που εκπονεί έναντι της, της, ε, του, του πληθυσμού του. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω ποιος είναι ο στόχος που θέλουμε να επιτύχουν αυτές οι κυρώσεις που επιβάλλουμε. Και παρακαλώ να μου το εξηγήσετε λεπτομερώς αυτό. Κλείνοντας, να πω ότι αυτά που είπε η κυρία Λοχπίλερ ε, τα ε, συμφωνώ, είναι σημαντικά. Ε, να έχουμε μια συγκεκριμένη θέση ε, των Ευρωπαίων πολιτών έναντι των πολιτών μια τόσο μεγάλη χώρα όπω είναι το Ιράν. Γιατί πραγματικά είναι τελείω διαφορετική η κατάσταση ε, με τα μάτια των πολιτών. Πρέπει να δούμε λοιπόν και εμείς ποια είναι η άποψη των πολιτών του Ιράν, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τα κατάλληλα μέσα για να τους εξυπηρετήσουμε, για να τους βοηθήσουμε. Να επιβάλλουμε μόνο κυρώσεις και να δείχνουμε μόνο τη δύναμή μας ποτέ δεν έχει δείξει ε, καλά αποτελέσματα και δεν έχει αλλάξει την κατάσταση. Ευχαριστώ. Grazie, collega Lösing. La parola al... Μάλιστα, το λόγο έχει ο κύριος ε, Αρλάκη. Βλέπω ότι υπάρχει σχετικά μεγάλη συνένεση για το γεγονός ότι αυτή η έκθεση είναι ατελής και έχει ε, ελλειπή ισορροπία και επίσης δεν συμβάλλει στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής πολιτικής απέναντι στο Ιράν, πράγμα το οποίο χρειαζόμαστε. Θα πρέπει να διορθωθεί Δεν ε, θα πρέπει να αρκεστούμε στο να επισφραγίσουμε την τελευταία θέση του State Department, να διαπιστώσουμε την κατάσταση, να ξεκινήσουμε από, την από το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει τα δικά της συμφέροντα και πολιτική απέναντι στο Ιράκ. Δεν μπορούμε απλά να επαναλαμβάνουμε αυτά που λέει τώρα το State Department σε αντίφαση στον... στα όσα είχε πει πριν από 4-5 μήνες σε πολύ κρίσιμα ζητήματα του πυρηνικού φακέλου. Συμφωνώ λοιπόν με τη θέση της συναδέλφου Λόκμπερ και Μονής Δερκίζα, διότι όντως μίλησαν για την περιπλοκότητα της κατάστασης και ελπίζω πως οι τροπολογίες θα διορθώσουν τον τόνο και τη θέση αυτής της έκθεσης. Τα δύο κύρια θέματα είναι η έλλειψη διάκρισης ανάμεσα στο Ιράν υπό το σημερινό καθεστώς και το Ιρανικού λαού από την άλλη πλευρά. Ο Ιρανικός λαός είναι ένας από τους πιο πολιτισμένους, προηγμένους και δημοκρατικούς λαούς του κόσμου. Αν ήταν ελεύθεροι να εκφράζουν τις θέσεις τους, το Ιράν θα ήταν μια δημοκρατική χώρα όπως οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Οποιοςδήποτε γνωρίζει το Ιράν, ακόμα και από μακριά το γνωρίζει αυτό. Και θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι ο Ιρανικός λαός είναι πολύ περήφανος για τη χώρα του και ότι η πλειοψηφία του κόσμου, του Ιρανικού λαού, είναι μεταρρυθμιστές και δεν θα συμφωνούν, δεν συμφωνούν με τις ευρωπαϊκές και τις, και τις αμερικανικές πολιτικές, ιδιαίτερα στη χρήση των κυρώσεων. Οι κυρώσεις δεν μπορεί να είναι τυφλές, δεν μπορεί να χτυπούν τον Ιρανικό λαό. Γιατί αυτό που κάνουν τελικά είναι να ενισχύουν τον Αχμαντινεζάτ και το τρομερό το αυτό καθεστώς. Όλοι γνωρίζουν στον ΟΗΕ ότι οι μη ευφυείς κυρώσεις ενισχύουν αυτά τα πολιτικά καθεστώτα αντί να τα αποδυναμώνουν. Και αυτό συμβαίνει σήμερα και στο Ιράν. Κάποιοι μιλούν για ευφυείς κυρώσεις, ας πούμε κάποιες κυρώσεις ε, για τους ανθρώπους ε, που ανήκουν στους ε, επαναστατικούς Besides being a big damage to, to Europe, φρουρούς της Επανάστασης, κυρώσεις δηλαδή στοχοθετημένες εναντίον συγκεκριμένων μόνο καθεστώτων χωρίς δηλαδή να αποδυναμώνεται η πρόοδος της Ιρανικής Δημοκρατίας. Ε, τώρα, άλλη έλλειψη διάκρισης που υπάρχει σε αυτή την έκθεση είναι το πολιτικό θέμα, όπου δηλαδή εμείς οφείλουμε να έχουμε μια ισχυρή θέση και να αγωνιστούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να στηρίξουμε τη δημοκρατία στο Ιράν με κάθε δυνατό τρόπο και του πυρηνικού φακέλου. Αν τα συγχαίουμε αυτά τα δύο, δεν ε, κάνουμε κάτι ευφιές, βλάπτουμε για τα συμφέροντα της Ένωσης αντιθέτως. Διότι το να, απορρίπτουμε την ε, τουρκική και βραζιλιάνικη πρόταση όταν όλοι οι πυρογνώμονες, ακόμα και οι πιο καλοί Αμερικανοί πυρογνώμονες θεωρήσαν ότι ήταν μία λύση στο θέμα του πυρηνικού φάκελου, αυτό δεν συμβάλλει δεν συμβάλλει στην ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στο Ιράν. Η τουρκο-βραζιλιάνικη έκθεση αρχικά έγινε δεκτή από τον πρόεδρο Ομπάμα γιατί δεν έλεγε τίποτα άλλο. Στην ουσία επαναλάμβανε αυτά που πρότειναν οι Αμερικανοί τον Οκτώβριο του περσινού έτους. Ήταν πολύ, μια πολύ λογική και ευφύης πρόταση και θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να ευχαριστήσουμε τη Βραζιλία και την Τουρκία που κράτησαν αυτή την θέση, ότι, γιατί είναι ένας τρόπος να προχωρήσουμε και να αποφύγουμε την άλλη λύση. Κυρώσεις και τελικά πόλεμος. Ως Ευρωπαίοι που είμαστε ελληνικοί άνθρωποι, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει το κόμμα του πολέμου που, ε, που ενδυναμώνεται στην, στη ΣΥΠΑ ε, και τροφοδοτείται από τους ανθρώπους της ε, οπλοβιομηχανίας. Μετά από το Ιράκ και μετά από το Αφγανιστάν θέλουν κι άλλα. Θέλουν επικυρώσεις, το Ιράν το απεικονίζουν στο παραβάτη της διεθνής νομοθεσίας κτλ. κτλ όταν το Ιράν στο θέμα του εμπλουτισμού του Ιρανίου έχει απόλυτο δικαίωμα να το κάνει σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Και είναι πάρα πολύ ισχυρή η θέση αυτή και δεν εξαρτάται από τον Αχμαντίνεζα και το καθεστώς. Για αυτό το σημείο όλοι οι μεταρρυθμιστές στο Ιράν, όλοι οι άνθρωποι που τους εμείς υποστηρίζουμε συμφωνούν. Συμφωνούν. Διότι αυτό είναι ένα δικαίωμα του Ιράν. Η λύση λοιπόν θα πρέπει να αναζητηθεί σε άλλε προτάσει και η τουρκοβραζιλιάνικη πρόταση ήταν πολύ καλή. Τελευταίο τμήμα λοιπόν της έκθεσης που λέει ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να κατηγορήσουμε την, τουρκική κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στο Ιράν θα πρέπει να διαλάξει τελείως. Εγώ θα υποβάλω σχετικές τροπολογίες. Η Τουρκία συμβάλλει θετικά για τη διεθνή λύση ενός μεγάλου προβλήματος και το σημείο 23 που λέει «Καλή το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συντονίσουν τις πολιτικές τους προς το Ιράν με αυτή της Ουάσιγκτον είναι απόλυτος περιττή και πρέπει να αποφευχθεί στο τελικό κείμενο. Ελπίζω ότι ο συνάδελφος δεν θα θεωρήσει ότι είναι προσωπική επίθεση. γνωρίζω πάρα πολύ καλά το Ιράν γνωρίζω το μεταρρυθμιστικό κίνημα, έχω επισκεφθεί τη χώρα πανελειμμένος και πραγματικά μιλώ με μεγάλη συμπάθεια προς τη χώρα αυτή και ελπίζω να μπορέσω να συμβάλλω σε ένα καλύτερο Ιράν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος Λαντσμπέργης και μετά ο κύριος Αλαφράγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξετάζοντας ε, την ε, πλήρη και ισορροπημένη έκθεση του κυρίου Μπέλντερ, βλέπω ότι λείπει ένα σημαντικό θέμα στην προσέγγιση μας διεθνώς. Το θέμα της δημοκρατίας δεν αναφέρεται καν. Ήταν σωστή, ήταν σκόπιμο να πούμε δύο λόγια και γι' αυτό, γιατί εκεί που αναφέρεται η δημοκρατία του Ιράν θα πρέπει να αναφερθεί και κάτι περί δημοκρατίας και μία μικρή τροπο, τροπολογία. Είναι από τα πιο ανησυχητικά καθεστώτα από το, τις χώρες που δεν είναι δημοκρατικές. Υπάρχουν και άλλα αντιδημοκρατικά καθεστώτα, αλλά το πιο επικίνδυνο από όλα είναι το Ιράν. Ο κύριος Αλαφράγκα, ευχαριστώ. Θα ήθελα να εκφράσω συντομία τη γνώμη μου, γιατί τη γνώμη της ομάδας την παρουσίασε ο κύριος Γκάλερ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπέλντερ για το έργο που επιτέλεσε και νομίζω ότι η έκθεσή του αποτελεί μια εξαιρετική βάση για την σύνοψη της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όχι μόνο παραλαμβάνοντας τα προηγούμενα ψηφίσματα, αλλά δίνοντας και κάποιες μελλοντικές προοπτικές για τη σχέση μας με τη χώρα αυτή. Το Ιράν θα είναι σημαντικός παράγοντας ε, στην παγκόσμια σκηνή και όχι μόνο στη Μέση Ανατολή. Μπορούμε λοιπόν να διαπιστώσουμε ότι σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες ό,τι αφορά την παραβίαση εκ μέρους του Ιράν του, ε, της συνθήκης για τη μη διάδοση και μάλιστα η έκθεση της ε, Διεθνούς Οργάνωσης Ατομικής Ενέργειας ήταν σαφής και είναι σαφές γιατί το, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υπερψήφισε ε, τις ε, κυρώσεις κατά του Ιράν, ακόμη και χώρες που αρχικά ήταν απρόθυμες όπως η Κίνα και η Ρωσία. Αυτά λοιπόν είναι όλα συζητήσιμα. Αυτό όμως που δεν αμφισβητείται που δεν είναι, είναι η κατάφορη και αποτρόπια παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πραγματοποιεί η χώρα αυτή και δεν μπορούμε παρά να τις ε, τονίζουμε με σθένος. Και νομίζω ότι η πυγμή θα πρέπει να είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό της ε, πολιτικής μας προς το Ιράν. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς ε, με προηγούμενες αρχές που έχουμε εκφράσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να ζητούμε από έναν εισηγητή να φάσκει και να αντιφάσκει. Γιατί η μεν μιλούν για παραλήψεις, η δε για πλεονασμούς. Γι' αυτό υπάρχει διορία για τις ε, τροπολογίες, για να βρούμε κοινέ λύσεις και συμβαστικές προτάσεις και να δούμε αν θα καταλήξουμε σε μια προσέγγιση κοινή που θα ανταποκρίνεται σε ευαισθησίες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προς τη χώρα αυτή που είναι ε, σημαντική αιστεία αστάθειας αλλά και από τις σημαντικότερες μαύρες τρύπες της διεθνούς πολιτικής. Και η πολιτική της ε, συγκατάθεσης δεν νομίζω ότι θα αποφέρει καρπούς, της συγκατάβασης μάλλον. Ο κύριος Μπέλντερ ε, ήταν αρκετά μετριοπαθής, προσπάθησε με συμβαστικό πνεύμα να γεφυρώσει τα κενά μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Σίγουρα πολλά σημεία θα πρέπει να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω, αλλά δεν μπορούμε παρά να είμαστε ευγνώμονες προς τον κύριο Μπέλντερ για την έκθεσή του, το έργο του, την προθυμία του, και να εκμεταλλευτούμε τον υπόλοιπο χρόνο για να καταλήξουμε στις συμβαστικέ λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις ευαισθησίες μας. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω καμία άλλη παρέμβαση. Το λόγο έχει ο κύριος Μπέλτερ για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν ήταν στο χέρι μου πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, τότε θα είχα αποβάλει ένα κείμενο που θα ήταν τέσσερις φορές όσο είναι αυτό. Ε, χρειάστηκε πραγματικά να διαγράψω, να συμπτύξω τόσα πολλά πράγματα. Στην ανταλλαγή απόψεων αναφέρθηκε και το θέμα της, ε, του τι κάνουμε με το γυναικείο κίνημα. Είχε συμπεριληφθεί στο αρχικό κείμενο, αλλά έπρεπε δυστυχώς να αφήσω πολλά πράγματα εκτός της ε, έκθεσής μου γιατί δεν είχα τον χώρο. Καταλαβαίνετε. Ακούστηκε η, ε, όρος εμπάθεια από τον κύριο Αρλάκη. Ο κύριος Αρλάκη γνωρίζει πως έχει η κατάσταση, η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της χώρας, έχει πάει πολλές φορές και υπάρχουν 150.000 ε, άνθρωποι σπουδασμένοι με προσόντα οι οποίοι φεύγουν από τη χώρα, μεταναστεύουν γιατί δεν αντέχουν άλλο. Μιλούμε για αρκετά δηλαδή δισεκατομμύρια το χρόνο τα οποία ε, εκραίουν από τη χώρα. Νομίζω ότι είναι λίγο κοινική αυτή η παρατήρηση. Για την μεγάλη κατάχρηση των υποδομών, των πόρων της, ε, της χώρας. Εγώ πραγματικά συμμερίζομαι πάρα πολύ τον Ιρανικό λαό και ελπίζω κάποια στιγμή να βρεθεί ένα καθεστώς που θα είναι λίγο πιο ανθρώπινο προς αυτούς. Να μην παρεξηγηθώ. Θα, το, θα, θα κάνω και εγώ κάποιες αλλαγές στην ε, γνωμοδότησή μου και θα το αναφέρω. Ε, τώρα, και εμένα με εντυπωσίασε ο τρόπος με τον, με τον οποίο τον... Ε, ο πρόεδρος ε, πραγματικά ε, επικρίθηκε από τους υπόλοιπους ε, για την ε, δημιουργία της κυβέρνησής του. Ε, είναι ενδιαφέρον όμως που βλέπουμε ότι υπάρχουν και στο εσωτερικό της χώρας πολλές και διαφορετικές απόψεις. Και είναι επίσης σημαντικό να δούμε ποιες είναι και οι θρησκευτικές πεπιθήσεις που υπερισχύουν. Επίσης αυτό που είπε ο συνάδελφος από τους σοσιαλιστές. Μιλούμε για μια Ισλαμική πολιτική με μεγάλη όμως σουνητική μειοψηφία. Δείτε και την περίπτωση Αστιάνη. Και αυτό είναι κομμάτι του προβλήματος. Ε, το θέμα των, των λιθοβολισμών. Ε, στις εφημερίδες πριν από λίγο καιρό υπήρχε και ένα πολύ ωραίο άρθρο για το θέμα αυτό. Θα προσπαθήσω λοιπόν, θα προσπαθήσω πραγματικά με τις τροπολογίες να καταστήσω πιο σαφές το πώς μπορεί κανείς εκ των έσω να ενισχύσει, να παρέμβει στην κατάσταση και να βοηθήσει τη χώρα. Η εσωτερική κατάσταση είναι πραγματικά πάρα πολύ περίπλοκη. Μπορώ να σας πω πολλά πράγματα. Ε, απόψεις δηλαδή από διάφορους επιστήμονες ανεξάρτητους ε, που το αποδεικνύουν αυτό, ότι πραγματικά ε, πρέπει να υπάρχουν ε, ειδικοί που αναλύουν την κατάσταση στο Ιράν, γιατί είναι πολύ περίπλοκη. Φυσικά πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία διαθέσιμα. Και ένα εξ αυτών έχει να κάνει με την επαναστατική φρουρά η οποία έχει επιβάλει μια μεγάλη οικονομική ιδιωτικοποίηση. Γι' αυτό καταλήξαμε σε αυτό το σλόγγαν ε, που είναι τα λεφτά από τα πετρέλαια. Ε, τώρα, για την εσωτερική ε, κατάσταση και τα ανθρώπινα δικαιώματα Εκεί βέβαια υπάρχουν πολλά να, να πούμε. Φυσικά υπάρχουν πολύ περισσότερα που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην έκθεση. Υπάρχουν ε, πραγματικά κατάφορες παραβιάσεις ανθρωπινών δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε απλώς στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι να κάνουν. Πρέπει και εμείς να δραστηριοποιηθούμε. και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμβάλλει με το δικό του τρόπο. Για την ε, πυρηνική ενέργεια και το σχετικό κεφάλαιο φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα αυτό. Απ' την άλλη όμως έχουμε και μια ευρωπαϊκή πολιτική που πρέπει να εφαρμοστεί. Μιλούμε για ε, κυρώσεις, λογικές κυρώσεις πάντα, ώστε να καταλήξουμε σε μια λύση. Ε, αυτό ίσως... και μάλλον κάτι που θα μπορούσε ίσως να, να είναι καλύτερο είναι να δούμε και τι γίνεται στον αραβικό κόσμο, όπου πολλές φωνές λένε ότι θα, αν συνεχίσει την πολιτική του το Ιράν θα καταλήξουμε δυστυχώς σε στρατιωτικές παρεμβάσεις. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα έχουμε υπόψη μας. Και κλείνοντας, για το ρόλο της Τουρκίας. Έχω πει ποια είναι η άποψή μου. Αν είχαμε το σχέδιο να μιλούμε για το Λίβανο και να του επιβάλλουμε κάτι, ότι να αυτό είναι προβοκάτσια, τότε είναι προφανές το τι κάνει το Ιράν για την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι και οικονομικοί βεβαίως αλλά αν κάποιος θέλει έτσι να ωρεοποιήσει την ε, τουρκική πολιτική εντάξει μπορεί να το κάνει απ' την άλλη όμως υπάρχουν ε, τεράστιες διαφορές απόψεων ε, μεταξύ των εμπλεκομένων. Εφόσον όμως μιλούμε για ευρωπαϊκή πολιτική η οποία υπάρχει, τότε θα πρέπει αυτή να εφαρμοστεί. Πάντα παραπονιόμαστε ότι δεν, υπάρχουν, ε, δεν ακολουθούν οι πράξεις τα λόγια μας. Ε, δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να μας ε, ε τυλίξει στο μικρό του δαχτυλάκι. Έχουμε και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου ασφαλεία. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει, υπάρχουν πολλά που πρέπει να συμπεριληφθούν εδώ. Αυτά από μένα πρόεδρε και ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Πρόεδρε, δεν ήθελα να πάρω το λόγο εγώ, αλλά ο Συνάδελφος ε, ε, Αρλάκη πήρε το λόγο από, για τη δική μας ομάδα, αλλά ε, αυτά που είπε ο συνάδελφος Μπέλντερ με έκανα να θέλω να πάρω το λόγο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να υιοθετήσει μόνο την, ως, ως θέση του την, τις θέσεις εδώ των των ε, μεμονωμένων βουλευτών. Πρέπει να έχουμε μια κοινή θέση, η οποία όμως να υποστηρίζεται από την πλειοψηφία. Ε, τα σχόλια των, ε, των συναδέλφων με κάνουν λίγο να διστάζω γιατί δεν νομίζω ότι αυτό το έχουμε κατανοήσει, το έχουμε χωνέψει ακόμα και δεν ξέρω κατά πόσο έχει βρει εφαρμογή και μέσα στην γνωμοδότηση. και για το Κοινοβούλιο θα ήταν άσχημο να υπάρχει ένα σχέδιο γνωμοδότησης για το Ιράν η οποία δεν θα εγκριθεί ή θα παραπεμφθεί πάλι πίσω στην Επιτροπή. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Αλλά θα μπορούσε να συμβεί. Αν δηλαδή ο εισηγητής δεν ε, λάβει υπόψη του τα σχόλια των, τις απόψεις των, ε, των ε, συναδέλφων που έχουν διαφορετική άποψη και βεβαίως δικαίως και καλά κάνουν και την έχουν. Με βάση την παρέμβαση του συναδέλφου να πω ότι η διορία για την υποβολή τροπολογιών είναι 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα και ψηφοφορία στην Επιτροπή 30 Νοεμβρίου 2010. Υπάρχουν μέσα για να μπορεί κανεί να παρέμβει στην έκθεση. Το λόγο, το τελευταίο, ο συνάδελφος Μπέλτερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να φοβάται η κυρία Νάιτς. Θα υποβληθούν τροπολογίες Οπότε φυσικά θα ληφθούν υπόψη οι απόψεις και μετά θα ψηφίσουμε. Οπότε θα αποφασίσουμε. Εγώ ευχαρίστως να λάβω σοβαρά υπόψη μου τις τροπολογίες σας και θα προσπαθήσω φυσικά να καταλήξω και σε κάποιες συμβαστικές προτάσεις. Δεν είναι αυτό, είναι εκ των ανουκάνευ. εφόσον βεβαίως υπάρχουν ε, ρεαλιστικά, πρακτικά επιχειρήματα. Δεν μπορούμε να μιλούμε με συναισθηματισμού σε μια έκθεση. Όταν θα υποβάλω κάτι, ε, ελπίζω να θα είναι μάλλον ε, πλήρες και από βιβλιογραφία και από μελέτη και από επιστημονικές ε, ε, αποδείξεις και από επιχειρηματολογία. Μην φοβάστε. Sorry. No, no, fait personnel, je m'excuse. Sull'ordine dei lavori? No. Για την ημερήσια διάταξη. Όχι, θέλω να απαντήσω στα όσα είπε ο συνάδελφο για σε προσωπικό επίπεδο. Εγώ ε, περιμένω την ίδια αντιμετώπιση από εσά με αυτή που είχα και εγώ για την ε, σύσταση της τελευταίας κυβέρνησης στην ε, Ολλανδία. Παρακαλώ να είσαστε λίγο πιο περιορισμένος όταν εκφράζεστε. εγώ θέλω να κλείσω εδώ τη συνεδρίαση. Έχει τελειώσει η συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Και θα τα πούμε το απόγευμα.